ε, την έκθεση του κυρίου Παρό για την ε, επιχειρησιακή ε, ευθύνη θα αναβληθεί κατά ένα μήνα ακολουθώντας την καθυστέρηση στην επί της ουσίας αρμόδια επιτροπή. Εάν δεν υπάρχουν άλλες παρατηρήσεις μπορεί να υιοθετηθεί η μερίσια διάταξη. Ευχαριστώ. Δεν υπάρχουν αντιρρήσεις ως προς τα πρακτικά. οι συντονιστές συμφώνησαν ε, να έχουν έκτακτη συνεδρίαση στις 17 Μαΐου για να εξεταστεί το σχέδιο έκθεσης για τις κατευθυντήρες γραμμές για την απασχόληση από τις 7 το βράδυ μέχρι τις 8.30 και θα ανακοινώσουμε αργότερα σε ποια αίθουσα θα πραγματοποιηθεί. Ε, διάσκεψη των Προέδρων 22 Απριλίου αποφασίστηκε να αναβληθεί η έγκριση ε, των ε, γενικών ε, κατευθυντηρίων γραμμών για την οικονομική πολιτική και την απασχόληση μέχρι να πληρούνται οι προϋποθέσεις για τη στρατηγική 2020. Οι συντονιστές λοιπόν συμφώνησαν να τροποποιήσουν το χρονοδιάγραμμα για την έγκριση της έκθεσης του κυρίου Ορή που προβλέπεται τώρα για τον, Απρίλιο, για τον Ιούλιο. Συγγνώμη. Επίσης θα βρείτε στο φάκελό σας ανακοίνωση σχετικά με ανταλλαγή απόψεων με ε, τον Επίτροπο για την ε, Στρατηγική 2020. Η ανακοίνωση υπάρχει στα δανέζικα αγγλικά, γερμανικά, συγγνώμη, αγγλικά και γαλλικά μόνο. Άλλο που έχετε στα φακέλους σας ε, αφορά την ανταλλαγή απόψεων με εκπροσώπους των κοινωνικών εταίρων και των μη κυβερνητικών οργανώσεων για την πρόσβαση των νέων στην αγορά εργασίας. Η πρώτη έκθεση που θα συζητήσουμε έχει να κάνει με την ενιαία, υποβολή, ενιαία διαδικασία υποβολή αίτηση για τη χορήγηση άδεια διαμονή και εργασία και δίνω αμέσω το λόγο στον κύριο Σέρκα. Ευχαριστώ πολύ κυρία, κυρία Πρόεδρε. Θέλαμε να υπενθυμίσουμε ότι αυτή η οδηγία βρίσκεται σε μια κατάσταση όπου η ευθύνη αυτής της ε, Επιτροπής ε, είναι κοινή με την Επιτροπή ΛΥΜΠΕ. Είναι η Επιτροπή ΛΥΜΠΕ η οποία ασχολείται με τα πιο ουσιώδη θέματα της οδηγίας, μια οδηγία που ε, που ασχολείται με τη χορήγηση μιας ενίας άδειας διαμονής και εργασίας για τους μετανάστες τρίτων χωρών που εισέρχονται νόμιμα σε μια χώρα και σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία. Και όπως είχαν εξαγγείλει τα προγράμματα τα οποία συνιστούν την προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης να συγκροτήσει μια ενιαία πολιτική μετανάστευσης, αυτοί οι νόμιμοι μετανάστες απολαμβάνουν ίσα δικαιώματα με τους, ε, εθνικού, με τους εργαζόμενους που είναι υπήκοοι αυτής της χώρας. Ε, είμαστε υποχρεωμένοι να συνεργαστούμε με την Επιτροπή ΛΥΜΠΕ και έχει γίνει μια μερασιά όπου η Επιτροπή ΛΥΜΠΕ ασχολείται κυρίως με τα νομικά θέματα της εμβέλειας της εν λόγω οδηγίας και όλα τα νομικά στοιχεία που σχετίζονται με το ε, χορήγηση μιας ενίας άδειας. Εμείς έχουμε κάποιες αρμοδιότητες σε σχέση με τα δικαιώματα και σε σχέση με την έκφραση των δικαιωμάτων που έχουν αυτοί οι εργαζόμενοι και επίσης με τους περιορισμούς των δικαιωμάτων σε ορισμένες χώρες ε, μέλη. Εγώ είχα την τύχη να έχω μια πολύ καλή συνεργασία εκ μέρου των άλλων εισηγητών και σήμερα βρισκόμαστε σε θέση να καταρτήσουμε μια πλατιά συνένεση σχεδόν ως προς το σύνολο των τροπολογιών που έχει κατατεθεί περιλαμβάνουν οι τροπολογίες αυτές σημαντικά θέματα, αλλά δεν έχουν οριστικό χαρακτήρα για όλες τις ομάδες και υπάρχουν και άλλα θέματα που άπτονται της πολιτικής μετανάστευσης και για τα οποία θα πρέπει να γίνει μια προσπάθεια από όλες τις πολιτικές ομάδες. Εγώ θα ήθελα να αναφερθώ κυρίως σε εκείνα τα θέματα που είναι πιο σημαντικά και που θα μπορούσαν να σηματοδοτούν μια πιο δυσχερή κατανόηση εκ μέρους ε, των ε, μελών. Αλλά ελπίζω ότι αύριο θα μπορέσουμε να υπερψηφίσουμε την έκθεση μια πλατιά, με μια μεγάλη πλειοψηφία. Ξεκινάμε με την ε, τροπολογία. Έχουμε μια τροπολογία υπαριθμών 24, δύο συναδέλφων από τη Φιλανδία, η οποία εισάγει μια συζήτηση που συνδέεται με ένα θέμα νομικής φύσεως ε, κατά πόσο μπορούν να γίνουν αποδεκτέ αυτές οι προτάσεις. Αυτές οι τροπολογίες προσπαθούν να εξαιρέσουν από τα δικαιώματα ε, ε, του εργαζόμενου που δεν έχουν μία σύμβαση και το θέμα αυτό με τον ε, τομέα εφαρμογής της οδηγίας. Θα ήθελα να, στήσω ποια, να ρωτήσω ποια είναι η γνώμη της νομικής υπηρεσίας, γιατί προσωπικά εγώ δεν νομίζω ότι μπορούμε να ψηφίσουμε σήμερα ε, θέματα τα οποία είναι αντικείμενο συζήτηση στην Επιτροπή ΛΥΜΠΕ. Εάν αυτή η τροπολογία δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή, κάθε αναφορά στις ε, συμβάσεις αυτές... Εγώ θα πρότεινα να να, να συνδέσουμε με την τροπολογία 24 την τροπολογία 9. Το δεύτερο θέμα που, προέλε, προήλθε από τη συζήτηση και με την Επιτροπή που μας έδωσε τη συνδρομή της είναι αυτό το οποίο συνδέεται με τους εργαζόμενους που υπάγονται στην οδηγία του 96 Σύμφωνα με το κείμενο της ε, Κομισιόν, αυτοί οι εργαζόμενοι που αποστέλλονται σε μια χώρα ε, της Ένωσης ε, εκτός της δικής σου, αυτοί οι οποίοι αποσπώνται δηλαδή σε μια άλλη χώρα, δεν έχουν ίση μεταχείριση. Έτσι λέει το κείμενο της οδηγίας. Και αυτό βεβαίως γύρει ένα θέμα νομικής ερμηνείας. Δεν έχουν ίση μεταχείριση με τους εργαζόμενους της χώρας υποδοχής ή διαρριγνύεται η αρχή της ίσης μεταχείρισης μεταξύ εργαζομένων που έχουν αποσπαστηθεί εφόσον προέρχονται από μια άλλη χώρα. Η Επιτροπή πάντοτε είπε στην νομοθετική πρωτοβουλία δεν ε, θέλει να επιβάλλει διακριτική μεταχείριση στους εργαζόμενους που αποσπώνται. Είτε είναι υπήκο μιας χώρας μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε είναι υπήκο μιας τρίτης χώρας. Η Επιτροπή μου απέστειλε μία, ένα κείμενο το οποίο θα μπορούσε τελικά να οδηγήσει σε μία λύση σε αυτό το θέμα ε, νομικής ε, φύσεως. Και που σχετίζεται βεβαίως και με την τροπολογία του κυρίου Τόμας Μαν υπαριθμών 25 που επίσης αναφέρεται σε αυτό το θέμα της απόσπασης των εργαζομένων. Εγώ ωστόσο θα ήμουν διατεθειμένος να παρουσιάσω ένα πακέτο ε, συμβιβασμών που να συμπεριλαμβάνει μια προφορική τροπολογία και να εισαγάγει μια νέα αιτιολογική σκέψη. Και ζήτησα από τη νομική υπηρεσία να μην ασχοληθεί, να μην αλλάξει η, οδηγία 26 και οι εργαζόμενοι εφόσον αποσπώνται να μην γίνονται αντικείμενο άνησης ε, μεταχείρισης. Αυτή είναι μια πρόταση που επέβαλα. Και εφόσον ε, λυθεί το θέμα αυτό, ο κύριος ε, Τόμας Μαν ε, μπορεί να διαγράψει το πρώτο τμήμα της τροπολογίας, το οποίο ακριβώς τα αυτού του θέματος. Το δεύτερο τμήμα της τροπολογίας του κυρίου Μαν ασχολείται με άλλα θέματα. Το τρίτο σημαντικό θέμα αφορά τους κανονισμούς για το συντανισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης που αφορά ένα εξαιρετικά πολύπλοκο νομικό σώμα που ρυθμίζει στην Ευρώπη τα δικαιώματα ενός εργαζόμενου ο οποίος εργάζεται σε πολλές χώρες. Και βεβαίω θα πρέπει να επιλύσουμε και το πρόβλημα των εργαζόμενων μέσω αυτή τη οδηγία που μετακινούνται σε διάφορες χώρες. Εάν θα έχουν ε, την ίδια μεταχείριση ή διαφορετική μεταχείριση από αυτό το σύστημα κανόνων που ακριβώς ορίζουν ε, συστήματα κοινωνικής ασφάλισης στη βάση ορισμένων εισφορών κλπ. Βάση μια ε, τεχνικής, πολύπλευσης τεχνικής που προβλέπει ο Ευρωπαϊκό Κοινοτικό κανονισμό. Υπάρχει εδώ ένα άρθρο και υπάρχουν αναφορές στις αιτιολογικές σκέψεις. Το ΕΛΚ έχει καταθέσει κάποιες τροπολογίες ε, και η ομάδα των Πρασίνων και εγώ ίδιος. Και συνεργαστήκαμε με την κυρία Ζιλ Λάμπερτ και σήμερα το πρωί εγώ ε, ε, συνεργάστηκα με την κυρία Όμεν Ρόιτερ, που είναι οι δύο πραγματικά εμπορευνόμενε σε αυτό το κοινοβουλίο σχέση με τον συντονισμό των συστημάτων αυτών και έχουμε μια συμβαστική τροπολογία που νομίζω μπορεί να τη ικανοποιήσει, η οποία απευθύνεται η οποία θα συμπληρωθεί τόσο στην αιτιολογική σκέψη όσο και στο ίδιο το κείμενο και θα ήταν ένα συμβασμός μεταξύ τριών τροπολογιών. Και ο συμβασμός τονίζει ότι αυτοί οι εργαζόμενοι θα έχουν τα δικαιώματα τα οποία έχουν αναγνωριστεί, τους αναγνωρίζονται σήμερα και αν αύριο ε, στο επίπεδο συντονισμού αυτών των ε, κανόνων βελτιωθεί αυτό το στάτους των εργαζόμενων, τότε οι εργαζόμενοι αυτοί θα έχουν το δικαίωμα να... Ε, θα μπορέσουν και αυτοί να βελτιώσουν τα δικαιώματά τους. Δεν πρόκειται δηλαδή να υπονομευθεί το, καθεστώς των δικαιωμάτων τους. Στην ε, οδηγία αυτή αναγνωρίζεται το δικαίωμα που έχουν οι εργαζόμενοι των τρίτων χωρών που έρχονται στις δικές μας χώρες μέλη και που έχουν τα δικαιώματα της κοινωνικής ασφάλισης. Και αυτό γύρισε ορισμένε χώρες μέλη και στην Επιτροπή ορισμένα προβλήματα ε, σε σχέση με ορισμένες πτυχές του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης. Και γι' αυτό υπήρξαν διάφορες τροπολογίες οι οποίες ε, προσπαθούν να ρυθμίσουν εντός εισαγωγικών το πρόβλημα ε, λέγοντας ότι κάθε χώρα μέλος ε, θα πρέπει να ρυθμίσει τα δικαιώματα της κοινωνικής ασφάλισης σε περίπτωση απόλυσης των επιδομάτων στην οικογένεια κλπ. Το σύνολο των κοινωνικών δικαιωμάτων. Και σε μια τροπολογία προβλέπει να αφαιθεί αυτό στην αρμοδιότητα των χωρών μελών το ρυθμίσουν όπως θέλουν. Αλλά στην περίπτωση αυτή, η οδηγία αυτή, κατά την άποψή μου, ε, θα έχανε απολύτω το νόημά τη γιατί θα υπήρχε καμία ισότητα στα δικαιώματα των εργαζομένων. Ωστόσο, υπάρχουν κάποιε χώρε μέλη που έχουν συστήματα κοινωνική ασφάλιση ιδιαίτερω πολύπλοκα και όπου τα δικαιώματα ε, εκχωρούνται όχι μόνο με το ε, δικαίωμα εργασίες αλλά με το δικαίωμα διαμονής. Και ε, τα δικαιώματα αυτά τα έχουν αυτή τη στιγμή οι εργαζόμενοι ε, φτάνουν σε μια χώρα, έχουν τα ίδια δικαιώματα όπως οι υπήκοοι αυτή τη χώρα. Και αυτό θέτει βεβαίω ορισμένα προβλήματα, γιατί δεν είναι φυσιολογικό κάποιο ο οποίο εργάζεται σε μια χώρα επί 30-40 χρόνια να έχει ακριβώ τα ίδια δικαιώματα με κάποιον ε, ο οποίο φτάνει από μια άλλη χώρα ευθύ εξ αρχή. Συνεπώ λοιπόν εδώ έχουμε τον συμβασμό γάμα όπου εκείνοι οι οποίοι θέλουν να εξαιρέσουν πλήρως τα δικαιώματα της κοινωνικής ασφάλισης από την ε, εμβέλεια της οδηγίας και να το αφήσουν στα ε, ευχέρια των κρατών μελών, αποδέχονται ένα συμβασμό ε, βάσει του οποίου γίνεται μια διάκριση μεταξύ δικαιωμάτων της κοινωνικής ασφάλισης τα οποία συνδέονται με τη χώρα διαμονής και τα δικαιώματα κοινωνικής ασφάλισης ε, που συνδέονται με την χώρα πρόλευσης των εργαζομένων. Και με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται ίση μεταχείριση. Όσον αφορά τα δικαιώματα κοινωνικής ε, ασφάλισης ε, που έχουν οι σε μία χώρα, μπορούν να περιλάβουν κάποια στοιχ... κάποιους όρους που συνδέονται ακριβώς με το καθεστώς διαμονής ενός εργαζόμενου σε μία χώρα. Αυτή είναι η τροπολογία που ζητήθηκε από κάποιες χώρες ε, λιγότερο πλούσιες που έχουν κάποια συστήματα επιδόματα και λοιπά, ε, επιδομάτων, βοηθημάτων κλπ. προς τις οικογένειες και ε, στην περίπτωση αυτή οι, οι χώρες αυτές συνδέουν τα δικαιώματα αυτά με το με την, με, το, με την άδεια διαμονής των εργαζόμενων και συνδέονται με κάποιες συγκεκριμένες προϋποθέσεις, αλλά με τον τρόπο αυτό δεν υποσκάπτεται η αρχή της ίσης μεταχείρισης. Αυτά, αγαπητοί συνάδελφοι, είναι τα πιο σημαντικά σημεία της συζήτησής μας. Οι υπόλοιπε ε, τροπολογίες ε, σε ορισμένα στοιχεία μας βρίσκουν σύμφωνους, αλλά όχι. Αλλά είναι λιγότερο σημαντικά θέματα και νομίζω ότι η αυριανή ψηφοφορία θα μπορέσει να είναι ε, συμβιβατή συμβατεί με διάφορες συμφορίες που έχουν γίνει στην δική μας Επιτροπή. Αλλά πιστεύω ότι θα πρέπει να ρυθμίσουμε αυτά τα τέσσερα σημεία τα οποία θα αποδώσουν στην έκθεση αυτή μια συνοχή ε, εξασφαλίζοντας την ίση μεταχείριση αλλά παρέχοντας ένα περιθώριο ευελιξίας σε ορισμένες ε, χώρες ε, μέλη όπου υπάρχει ανάγκη να ισχύσει η αρχή της επικουρικότητας. Uh, Σας ευχαριστώ πολύ. Πριν να δώσω το λόγο στην Τζιν Λάμπερτ, να πω ότι το θέμα που έθεσε σχετικά με την ε, μη ε, αποδοχή Η νομική υπηρεσία με ενημερώνει ότι αυτή η συγκεκριμένη τροπολογία δεν θα ψηφιστεί γιατί δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητές μας. Γι' αυτό και δεν θα την ψηφίσουμε. Η Τζιν Λάμπερτ. Ευχαριστώ και ευχαριστώ τον κύριο Σέρκας για την εισήγησή του. Τα θέματα που αφορούν την κοινωνική ασφάλιση. Να πω δύο λόγια από αυτόν. Οι τροπολογίε που εγώ κατέθεσα και οι συμβιβαστικέ τι οποίες τώρα φτάσαμε, στόχο έχουν να μην ε, περιχαρακώσουν την υφιστάμενη κατάσταση, ούτε να αποκλείσουν εξελίξεις για το μέλλον. Έχουμε ενημερώσει τον κανονισμό περί κοινωνικής ασφάλισης. Αν ε, και όσοι θέλουν να διατηρήσουν αυτή ε, την τυπική διαδικασία μπορούν να το σκεφτούν. Αν θέλουν δηλαδή να ακυρώσουν 10 χρόνια σκληρής δουλειάς. Πάντως, ούτως ή άλλως όλα αυτά δεν ε, έχουν στόχο να είναι τελείως άκαμπτα ως προς το μέλλον. Επίσης θα πρέπει να είναι σαφές πως ε, η πτυχή της κοινωνικής ασφάλισης, έτσι όπως εκτίθεται στον κανονισμό ή συντονισμός, σε πάση περιπτώσει, της κοινωνικής ασφάλισης, δεν αγγίζει τα επιδόματα προνοίας. Τα κράτη-μέλη είναι αυτά που είναι υπεύθυνα για αυτά. Δεν είναι η κλασική κοινωνική ασφάλιση όλα αυτά και αυτό θα πρέπει να το έχετε υπόψη όταν βλέπετε τις διάφορες τροπολογίες. Όσον αφορά την ε, συμπερίληψη των αποσπασμένων εργαζομένων, εγώ είμαι ευγνώμων για την ε, τροπολογία που κατέθεσε ο εισηγητής, γιατί νομίζω πως και αυτή βοηθά στο να αποσαφινιστούν ορισμένα από τα ζητήματα που προέκυψαν όσον αφορά την ενιαία άδεια. Ότι δηλαδή υπηκότητα των χωρών που έρχονται να εργαστούν. Προφανώς και συμπεριλαμβάνονται και η διατύπωση αυτή τώρα καθιστά απόλυτα σαφή τα δικαιώματά τους αν έρχονται ως αποσπασμένοι. Τι συμβιβαστικέ λοιπόν που έχουν κατατεθεί να τι υποστηρίξουμε και εν γέννη υποστηρίζουμε τη γραμμή που έχει ακολουθήσει ο εισηγητή. Σα ευχαριστώ. Η κυρία Όμενο Ρόιτεν. Μάλιστα, Πρόεδρε, είναι ε, μια πραγματικά πολύ δύσκολη υπόθεση, πολύ δύσκολο θέμα. Η Τζιν το γνωρίζει πάρα πολύ καλά, γιατί υπάρχει και ο συντονιστικός ε, κανονισμός, ο οποίος μας απασχόλησε για πολλά χρόνια. Και αυτή η νομοθεσία για τους εργαζόμενους τρίτων ε, χωρών έχει δώσει λαβή για διάφορες ερμηνείες. Περί τίνος πρόκειται. Πρόκειται για επικούς τρίτων χωρών που μπορούν να εργαστούν σε ένα κράτος μέλος της Ένωσης. Αυτό θέλουμε να ρυθμίσουμε. Και υπάρχουν και θέματα τα οποία δεν θέλουμε να τα ρυθμίσουμε και αυτό το λέω στον Μαν και σε άλλους υπάρχουν οι τον άσυλο, υπάρχουν οι φοιτητέ, αλλά αυτά δεν, αυτοί δεν εμπίπτουν σε αυτήν εδώ την οδηγία. Ας πούμε τα ε, οικογενειακά επιδόματα δεν έχουν ούτε και αυτά εδώ τίποτα να κάνουν. Δεν εμπίπτουν σε αυτή την οδηγία. Αυτά είναι τα πρώτα που ήθελα να πω, κυρία Πρόεδρε. Και έπειτα υπάρχει και ένα πρόβλημα το οποίο έφερνε και συνάδελφοι οι Φιλανδοί. Ο Αλεξάνδρος Σέρκας μας είπε πως είχε ρυθμιστεί το θέμα. Στη Φιλανδία όταν κανείς είναι φοιτητής έχει το δικαίωμα να εργαστεί κάποιες ώρες την εβδομάδα και χάρη σε αυτές τις κάποιες ώρες της εργασία μπορεί να έχει και πλεονεκτήματα που σχετίζονται με την εργασία και με την άδεια παραμονής στη χώρα. για τη Φιλανδία και για τι άλλε χώρες που εφαρμόζουν ένα τέτοιο σύστημα προσπαθήσαμε να βρούμε μια λύση και είπαμε ότι ε, θα πρέπει θα, η άδεια να δίνεται μόνο από τη στιγμή που έχουν εργασία και για τις όλε χώρες δεν θα πρέπει να τροποποιήσουν το σύστημά τους. Θα μπορούν δηλαδή να υπάρξουν κάποιες εξαιρέσεις για τα κοινωνικά ε, πλεονεκτήματα όταν ε, Αυτά συνδέονται με την άδεια παραμονής. Και έτσι λύσαμε το θέμα τη Φιλανδία. Και την περασμένη Πέμπτη έγινε μια συνεδρίαση και εγώ προσπάθησα να βρω μια κάποια λύση. Αν ήμουν, ας πούμε ότι ο Τόμας παντρεύεται μια πανέμορφη Βραζιλιάνα και αυτή ανέκαθεν είχε μια πολύ ενδιαφέρουσα δουλειά και θέλει να εργαστεί σε ένα, νοσοκομείο στο Μάστριχτ. Καταρχήν θα πρέπει αυτή η όμορφη κοπέλα να προσκληθεί από τις κάτω χώρες, γιατί διαφορετικά δεν θα μπορεί να εργαστεί στο εξωτερικό. Πρέπει να λάβει την άδεια εργασία της και στη συνέχεια να έχει και τα ωφέλη τα πλονεκτήματα που θα της δίνει αυτή εδώ η οδηγία. Στη συνέχεια, αν αποκτήσετε και ένα παιδί με αυτή την ε, κυρία, ο οποίο δεν είναι φοιτητή, δεν θα μπορεί να εκμεταλλευτεί αυτή εδώ την οδηγία. Μόνο αυτοί οι οποίοι έχουν έρθει για να εργαστούν ε, θα χαίρουν των ωφελών αυτή εδώ τη οδηγία. Δηλαδή πρόκειται για αυτού που έχουν προσκληθεί για να εργαστούν. Και έπειτα για του αποσπασμένου ε, ε, εργαζόμενου. Άκουσα πολύ καλά τον Αλεχάνδρο και τα όσα μα είπε. Και εγώ έχω την εντύπωση πώ είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Αλλά λέει, αν υπάρξει μια ας πούμε ισπανική εταιρεία που στέλνει έναν Ισπανό εργαζόμενο στι κάτω χώρε για να δουλέψει και έναν Βραζιλιάνο εργαζόμενο να δουλέψει, θα έχουν τα ίδια δικαιώματα. ο Βραζιλιάνος θα έχει, ανάγκη από άδεια εργασία. Πάντω. Ε, δεν ξέρω, ε, είναι κάπως μπερδεμένο το πράγμα όσον αφορά την ερμηνεία της απόσπαση. Νομίζω λοιπόν πως έχουμε έναν, ε, μια διατύπωση αρκετά αόριστη Τώρα, για τις ε, υποτροφίες. Νομίζω πως και εδώ θα πρέπει κάπως να τροποποιήσουμε τη διατύπωση για να μπορούν να ωφεληθούν κάποιοι υπότροφοι, αλλά για, κατά την άποψή μας δεν εμπίπτουν στο πλαίσιο αυτής της οδηγίας. Και έπειτα υπάρχει και το δικαίωμα στη σύνταξη αν κάποιος εργαζόμενος έχει μείνει πολλά χρόνια για να δουλέψει, θα πρέπει να έχει δικαίωμα στη σύνταξη, ακόμα και αν επιστρέψει στη χώρα του. Αν δούμε λοιπόν τις τροπολογίες 19 και 21, Έχουμε καταργήσει το 8, 5 και 9. για να γίνουν κάπως πιο ε, συνεπή τα πράγματα. Υπήρχε μια εξαίρεση για την Αυστρία και για τη Γερμανία, αλλά αυτή εξαφανίστηκε. Νομίζω πως ε, δεν θα υπάρχει λοιπόν πρόβλημα ως προς αυτό, αλλά εγώ θα ήθελα να ζητήσω από τον Αλεχάνδρο και τους συναδέλφους να ε, υποστηρίξουν τις τροπολογίες 29 και 21. Ευχαριστώ. Yes, thank you. Uh, Ευχαριστώ πολύ ο Τόμας Μάν. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Η ιδέα της Συρία με τη Βραζιλιάνα μου άρεσε πολύ. Ε, δεν ξέρω αν εννοούσε τον James Bond. Ε, αν ερχόταν η ωραία Βραζιλιάνα σε εσά ε, στην Ολλανδία θα έπρεπε να έρθει σε επαφή με τον κύριο Φανίστελ Ρόι. Ε, εν πάση Να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Εν πάση Αν έχουμε φοιτήτρια και υπάρχει κάποιο υπεύθυνο σε κάποια χώρα. Στην περίπτωση αυτή δεν είναι πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα, αλλά στην ε, τροπολογία 21 ε, που Ε, αναφέρομαι στην ε, οδηγία 859 κάθετος 2003. Δεν θα μπορούσαμε να έχουμε άλλες σοβαρές περιπτώσεις. Η οδηγία αυτή Εάν έχουμε κάποιον που εξαιρείται από την ε, οδηγία και έχει άδεια παραμονή. τότε μέχρι στιγμής έχει ερμηνευθεί ως εξή ότι θα δικαιούται κάποιες επιδοτήσεις όπως είναι για παράδειγμα επιδόμα, κάποια επιδόματα ε, για, για τα παιδιά του ή, ή αλλά επιδόματα τα οποία λαμβάνει κανείς στα πλαίσια μιας παραμονής στην ε, Γερμανία. Γι' αυτό η Γερμανία μέχρι τώρα είχε ένα σύστημα αδειοδότησης και γι' αυτό δεν μας αρέσει που στην ε, τροπολογία 21 που λέμε ότι θα πρέπει να ε, εξαιρέσουμε τις περιπτώσεις αυτές. Δεύτερη παρατήρηση, ο συνάδελφος ε, Τσέρκας στην τροπολογία 25 την έχει συμπεριλάβει σε μεγάλο βαθμό. Διαβάζω στα αγγλικά το δεύτερο μέρος. Λέει ότι δεν θίγει την αρμοδιότητα των κρατών μελών όσον αφορά την πρόσβαση και την εισδοχή υπηκών τρίτων χωρών στην αγορά εργασίας τους. Νομίζω ότι είναι πολύ ακριβή η διατύπωση αυτή και αυτό συνάδει με αυτό που είπε ο, ο, πριν ο συνάδελφο ε, Τσέρκα, ότι από τη μία έχουμε το δίκαιο που αφορά την παραμονή και το δίκαιο που αφορά την ε, απασχόληση. Αυτά θα πρέπει να τα διακρίνουμε. Χαίρομαι λοιπόν που έχει συμπεριλάβει την. Ε, τροπολογία υπαριθμών 25, τουλάχιστον το δεύτερο μέρο, που είναι και το σημαντικό. Και έχω μία ερώτηση. Ο συνάδελφο Τσέρκα είπε ότι μπορεί να υπάρξουν ακόμα κάποιοι συμβιβασμοί. Ίσως τώρα θα ήταν η ευκαιρία να ε, δούμε τις ε, τροπολογίες ε, έστω και στα αγγλικά ε, θα πρέπει να εξετάσουμε τις ε, αποχρώσεις στις ε, συμβιβαστικές τροπολογίες, διότι δεν μας ενδιαφέρει η γενική δήλωση, μας ενδιαφέρουν οι λεπτομέρειες οι οποίες, τις οποίες μπορούμε να κρίνουμε μόνο όταν τις δούμε στην στην αρχική γλώσσα. Θα παρακαλούσα λοιπόν τον κύριο Σέρκας να μου εξηγήσει λεπτομερώς σε κάποια ζητήματα, διότι μπορεί να καταλήξουμε σε άλλα ε, ε, αποτελέσματα από αυτά ε, στα οποία καταλήξαμε στις πολιτικές μας ομάδες. Κυρία Πρόεδρε, σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες όπως είναι η Φιλανδία, πραγματοποιείται μια έντονη συζήτηση για την μετανάστευση και γι' αυτό περιμένουμε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να έχουμε κανόνες για τη μετανάστευση, κοινούς κανόνες. Η πρόταση που εξετάζουμε αυτή τη στιγμή είναι θετική. Και θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Αλεξάνδρου Τσέρκας για την ευέλικτη στάση του όσον αφορά τα προγράμματα της Φιλανδίας. Όσον αφορά δηλαδή το γεγονός ότι το δικό μας σύστημα κοινωνικής πρόνοιας διαφέρει από τα συστήματα άλλων κρατών μελών και θα θέλαμε να διασφαλίσουμε την ίση μεταχείριση των ανθρώπων που έρχονται να εργαστούν στη χώρα μας. Είναι πολύ θετικό το θέμα αυτό και πρόκειται για τρόπο να προωθήσουμε τη μετανάστευση που θα βασίζεται στην απασχόληση. Αυτό είναι πολύ σημαντικό στην Ευρώπη λόγω της δημογραφικής κατάστασης. Ταυτόχρονα θα μπορέσουμε έτσι να εξαλείψουμε τα προβλήματα που μπορούν να προκύψουν. Για παράδειγμα, την κατάχρηση των εργαζομένων, την κακομεταχείρισή τους. Ε, πρόκειται για καλό σημείο κίνηση όσον αφορά τους αποσπασμένους εργαζομένους. Ε, περιμένω να δω τις τροποποιήσεις ε, στην οδηγία που αφορούν τους αποσπασμένους ε, εργαζομένους, ώστε να δούμε ακόμα καλύτερο αποτέλεσμα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την επιτυχή του έκθεση και είμαι βεβαία ότι οι πολίτες μας θα επικροτήσουν την έκθεση αυτή. Είναι γεγονός ότι επί 400 χρόνια οι Ευρωπαίοι εγκατέλειπαν την Ευρώπη σε αναζήτηση μιας καλύτερης ζωής. Ενώ τώρα η Ευρώπη προσελκύει ανθρώπους λόγω της σταθερότητας και του υψηλού βιωτικού επίπεδου. Γι' αυτό έχουμε τέτοιους κανόνες αυτή τη στιγμή. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Σέρκας για την ευέλικτη στάση του. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πιστεύω ότι το βασικό πρόβλημα με αυτήν την πρόταση είναι ότι ορισμένες ομάδες ανθρώπων ε, εξαιρούνται, αποκλείονται μάλλον από το φάσμα εφαρμογής, από το πεδίο εφαρμογής και από τις εξαιρέσεις. Είναι πολύ σημαντικό όλοι οι υπηκόοι των χωρών που νομίμως εργάζονται στην Ευρώπη να την χάνουν ίσης μεταχείρισης με τους πολίτες της Ένωσης, ε, τόσο στον κόσμο της εργασίας όσο και στο κοινωνικο-οικονομικό πλαίσιο. Όμως, οι εποχιακοί εργαζόμενοι, οι πρόσφυγες και οι αυτοπασχολούμενοι αποκλείονται από το πεδίο εφαρμογή τότε τη οδηγίες. Η Κομισιόν ενημέρωσε ότι το, την το καλοκαίρι θα δημοσίευε μια διαφορετική πρόταση οδηγία για τους εποχιακούς. Δυστυχώ, δεν είναι σαφές πότε θα αρχίσει να ισχύει αυτή η χωριστή οδηγία. Κατά την άποψή μου είναι απαραίτητο να συμπεριληφθούν οι εποχιακοί εργαζόμενοι σε αυτήν εδώ την οδηγία. Γιατί ο αποκλεισμό τους ε, ε, δεν είναι σωστός ο αποκλεισμό αυτός, ιδιαίτερα όσον αφορά σχετικά θέματα όπως οι συνθήκες εργασίας και το δικαίωμα του συνδικαλισμού. Οι εποχιακοί εργαζόμενοι να αποκλειστούν λοιπόν από αυτήν την οδηγία θα κινδυνεύουν να γίνουν αντικείμενα εκμετάλλευσης. Ευχαριστώ. Σα ευχαριστώ. Πριν να δώσω και πάλι το λόγο στον κύριο Σέρκα, θα πρέπει να έχουμε στο νου μα ότι έχουμε ακόμα πέντε λεπτά για το θέμα αυτό πριν μπούμε στο επόμενο. Ε, Μία σύντομη ερώτηση. Είπατε ότι θα προσπαθήσετε να βρείτε μια ισορροπία ανάμεσα στι δύο πλευρέ για την κοινωνική ασφάλιση και τα επιδόματα. Για την 22 δεν έχετε σημειώσει ποια είναι η θέση σας. Γιατί, όπως την ξαναείδα, φαίνεται ότι αφορά κάποια από τα θέματα για τα οποία μιλήσατε, κύριε Σέρκας. Sí, y empiezo por usted, señora presidenta, para decirle que en mi lista de voto la enmienda 22 está eh, aprobada en parte. Voy a pedir un split vote, de tal manera que voy a aprobar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 toma en consideración las enmiendas diecinueve y veintiuno de una manera armónica. Eh, Thomas Mann. Thomas Mann, ευχαριστώ πολύ που δεχθήκατε τη συμβαστική μου λύση σε σχέση με τροπολογία υπαριθμών 25 και θα ήθελα να σας ε, διαβάσω εντάχει τις συμβαστικές τροπολογίες αυτές οι συμβιστικές τροπολογίες δεν μπορούν να διαμεθούν αν δεν συμφωνήσουν οι συνάδελφοι. Αλλά όπως μου είπες ότι συμφωνείς ε, θα αποτελέσει το συμβιβασμό. Θα αποτελέσει το συμβιβασμό που αφορά τους ε, αποσπασμένους εργαζόμενους ε, και στη δική μου τροπολογία ε, συμπεριλαμβάνω όλες τις ε, προτάσεις της Επιτροπής και θα έλεγα το εξή. Οι υπήκοοι τρίτων χωρών που είναι αποσπασμένοι δεν καλύπτονται από αυτή την οδηγία. Αυτό δεν θα εμποδίσει τις ε, χώρες προέλευσης να αντισφυκώς ε, να, απολαμβάνουν στις χώρες ε, προέλευσης τα ίδια δικαιώματα ε, και στις χώρες όπου αποσπώνται. Να επηρεάζονται από την Οδηγία Περιεργαζομένων 9671. Ναι, είναι σαφές ότι εδώ δεν περιλαμβάνονται οι εργαζόμενοι οι οποίοι είναι αποσπασμένοι, αλλά ενώ αποσπώνται οι εργαζόμενοι αυτοί θα έχουν ίσα δικαιώματα ανεξάρτητα από την θαγένεια που έχουν ορισμένοι από αυτούς τους αποσπασμένους εργαζόμενους. Και αφήνοντας κατά μέρος ε, τις ε, σχέσεις με τη χώρα υποδοχής. Ε, εγώ εγώ θα ήθελα να αλλάξει η οδηγία αυτή, αλλά δεν είναι αυτή η ενδειγμένη στιγμή. Αλλά δεν θα ήθελα να ερμηνευθεί η εξαίρεση αυτών των εργαζομένων για να προσθεθεί μια νέα διακριτική μεταχείριση για τους εργαζόμενους που αποσπώνται. Η άλλη τροπολογία θα ήταν, είναι ο συμβασμός Β, ο οποίος ε, σχετίζεται με, τους, με τις διατάξεις για την κοινωνική ασφάλιση που έχουν ζητήσει οι βόρειες χώρες και οι Φιλανδοί και η οποία είναι ένα συμβασμός με τροπολογία 37-13 και την 36 του Γκουε, εφόσον η Γκουε συμφωνεί. Και εισάγει στο άρθρο 10 σημείο 2 ε, παράγραφος ε την εξής ε, διατύπωση. Τη διαβάζω αργά στα κακά μου αγγλικά. Μπορεί να περιορίσει την ίση μεταχείριση με τους ε, υπηκόους ε, της χρησιμοποιώντας τη λογικά κριτήρια παραμονής όσον αφορά τα, διάφορα επιδόματα, αλλά όχι τα επιδόματα απασχόλησης. Αν η άδεια είναι για διαφορετική χώρα ε, από αυτήν που είναι η άδεια της εργασίας. Συνεπώς μπορούν να θεσπιστούν διαφορετικά κριτήρια πιο περιοριστικά. Αλλά αλλά αφορούν τα επιδόματα τα οποία σχετίζονται με τη διαμονή και όχι τα επιδόματα που σχετίζονται με την εργασία. Τώρα, ο, ο συμβιβασμό Γ είναι η τροπολογία τη κυρία Όμεν Ρόιτερ και τη Jill Λάμπερτ που βασικά αφορά την 16 και 17, τη συμπεριλαμβάνει και εξαιρεί ε, ε, τις ε, παραγράφους 7, ε, 8 κλπ. Ευχαριστώ πάρα πολύ και θα ευχαριστήσω και την Λίζα και την γενεδορία της. Και θα ήθελα να πω ότι όλη αυτή η συζήτηση για τη μετανάστευση δεν θα πρέπει να μας κάνει να ξεχνάμε ότι μιλάμε για μια υπόσχεση που δώσαμε σε εργαζόμενους από άλλες χώρες ότι θα την χάνουν ίσης μεταχείρισης στην Ευρώπη Συνεπώς, το βασικό μας, ο βασικό μας γνώμονας θα πρέπει να είναι το κριτήριο της ίσης μεταχείρισης και η διαχείριση των δικαιωμάτων θα πρέπει να είναι δίκαιη. Αυτό προσπαθώ να κάνω εδώ. Εγώ συμμερίζομαι την ιδέα ότι οι εποχιακά εργαζόμενοι έως ότου έχουν μια δική τους κατάλληλη οδηγία θα πρέπει να συμπεριληφθούν σε αυτή την οδηγία. Γι' αυτό αναφέρεται στην αιτιολογική σκέψη ότι έχει έναν οριζόντιο χαρακτήρα. Αλλά ε, ελπίζω, το, ε, αλλά αυτό δεν είναι δική μας υπόθεση, ελπίζω ότι η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών θα υιοθετήσει αυτή την άποψη, θα υιοθετήσει αυτό το κριτήριο έως ότου, όπως σας είπα, ε, υπάρχει σερπιστή μια ξεχωριστή οδηγία για τους εποχιακά εργαζόμενους. Αλλά ελπίζω ότι θα γίνουν σεβαστά των εργαζόμενων αυτών. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Σάι ήθελε να παρέμβει, αλλά είχα κλείσει τον κατάλογο και έδωσα πάλι τον λόγο στον εισηγητή. Εκτό αν ε, θέλετε μια διευκρίνηση, ότι έχουμε μόνο 15 λεπτά για το επόμενο θέμα. Μπορείτε να το συζητήσετε αργότερα με τον κύριο Σέρκα. Ναι, ναι, μπορώ να το κάνω αν δεν έχουμε πολύ χρόνο. Ναι, μια διευκρίνηση, πολύ σύντομα. Ναι, μια προφορική τροπολογία. Όσον αφορά την προφορική τροπολογία τον περιορισμό αυτό που θα βασίζεται στην διαμονή ε, θα το συμπεριλάβετε και στην ε, προφορική τροπολογία. Uh, I think that it be there. Διότι πιστεύω ότι θα πρέπει να συμπεριληφθεί. Εάν αυτός ο περιορισμός που θα βασίζεται στη διαμονή, στην, παραμονή, πιστεύω θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται και στην προφορική τροπολογία ο περιορισμός αυτός. Κύριε Σέρκας. Ναι, κατά πάσα πιθανότητα ε, ε, ε, είναι δύσκολο να το... γιατί μιλάμε σε διαφορετικές γλώσσες, αλλά η δική μου προφορική τροπολογία αφορά την αιτιολογική σκέψη 12 και εκεί αναφέρεται στους αποσπασμένους. Δεν σχετίζεται με τους διαμένοντες. Είναι κατά πόσο εξαιρούνται ή δεν εξαιρούνται από την οδηγία οι αποσπασμένοι και η συζήτηση σχετίζεται με την ερμηνεία τι σημαίνει αυτή η εξαίρεση. Αλλά η διαμονή εδώ δεν παίζει κανένα ρόλο. Ε, στο άρθρο 12 αναφέρεται η... Ε, αναφέρεται ε, αλλά όχι στην ιδεολογική σκέψη 12 η διαμονή και πρόκειται για τα επιδόματα τα οποία συνδέονται με την διαμονή και για τα επιδόματα τα οποία συνδέονται με την εργασία. Στο άρθρο 12 εκχωρεί τη δυνατότητα στις χώρες μέλη να θεσπίσουν κάποια κριτήρια διάκρισης για τους μετανάστες όσον αφορά τα επιδόματα τα οποία σχετίζονται με, τα, με την διαμονή. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Η ψηφοφορία θα είναι αύριο στις 12 ε, η ώρα. Η Γκαμπριέλε Τσίμερ έχει το λόγο για την ε, έκθεσή της σχετικά με τη μείωση της ένδυας, δημιουργία θέσεων απασχόλησης, αναψώμενες χώρες κλπ. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλα τα μέλη της Επιτροπής, όλους τους συναδέλφους ε, που συμμετείχαν με την υποβολή τροπολογιών τους ε, στην έκθεση για τη μείωση της ένδυας ε, για την οποία η Επιτροπή μας γνωμοδοτεί. Γενικά βλέπω από τις τροπολογίες ότι γενικά στοχεύουν στις ε, αξιοπρεπείς θέσεις εργασίας καθώς και στην ανάπτυξη, κυρίως στην οικονομική ανάπτυξη η οποία θα πρέπει να συνδέεται με κριτήρια ανάπτυξης και δεν θα πρέπει να εξετάζεται ε, μεμονωμένα. Πιστεύω ότι αν μπορέσουμε τελικά να ε, συνδυάσουμε, να συντονίσουμε τις τροπολογίες, ε, θα ε, μπορέσουμε να έχουμε μια καλή θέση η οποία θα βελτιώσει την θέση της αρμόδιας επι... της ουσίας Επιτροπής Ανάπτυξης. Γι' αυτό θα ήθελα να πω ότι θα συμφωνήσω με όλες τις τροπολογίες ε, τις έχω εξετάσει, βρίσκω ότι ε, ταιριάζουν με το κείμενο και πιστεύω ότι αποτελούν λογική συμπλήρωση της έκθεσης ε, πριν κάποιους μήνες στην Επιτροπή Ανάπτυξης συζητήθηκε το θέμα του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας και πιστεύω, σε, ακρόαση και πιστεύω ότι είναι χρήσιμο εμείς ως Επιτροπή Απασχόλησης να προσπαθήσουμε εκ των υστέρων να συμπεριλάβουμε τις πτυχές που συζητήθηκαν τότε και πιστεύω ότι με τις τροπολογίες μας θα μπορέσουμε να ακουστούμε στην Επιτροπή Ανάπτυξης σε μία έκκληση κλείνοντας Κατά την εξέταση των μεταφράσεων παρακαλώ να ξεκινήσετε με βάση το αγγλικό κείμενο. Στο γερμανικό κείμενο βλέπω κάποιες ανακρίβειες, κάποια ερωτηματικά. Θα παρακαλούσα την γραμματεία να συνομιλήσει με την μεταφραστική υπηρεσία πριν την οριστική ε, υιοθέτηση του κειμένου μας. Θα ήθελα δηλαδή να φροντίσουν το και το γερμανικό κείμενο να είναι σωστό, να μην περιλαμβάνει λάθη. Επάσε τόσο η σημείο κίνησής μας είναι το αγγλικό κείμενο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ η κυρία Ντέβα. Ευχαριστώ πολύ κυρία Τσίμερ για αυτή την εξαιρετική εργασία και πραγματικά ήταν Χαρά μου που ασχολήθηκα με αυτή την έκθεση. Ωστόσο θα ήθελα να έχω δύο διευκρινήσεις. Καταρχήν η τροπολογία 12 που παρουσιάστηκε από την κυρία Γκρινή. Και σε ευχαριστώ πολύ για την τροπολογία αυτή που υπενθυμίζει ακριβώς την ανάγκη παρακολούθησης των νέων που τελειώνουν το σχολείο. Κάτι που τείνουμε να ξεχνάμε. Θα μπορούσατε όμως να μου διευκρινίσετε τι καταλαβαίνετε όταν λέτε την εφαρμογή κάποιων στάζ ποιότητας, υψηλής ποιότητας. Ε, αυτά τα στάζ θα είναι αμοιβόμενα, ε, θα είναι στο πλαίσιο του πανεπιστημίου. Αυτή είναι μια πρώτη ερώτηση. Και κυρία Τσίμερ, αν μπορείτε να μου διευκρινίσετε τι εννοείτε στην ε, τροπολογία υπαριθμών 25. Τι καταλαβαίνετε όταν λέτε ότι το Κοινοβούλιο και οι χώρες μέλη ελέγχουν τις ε, δυνατότητες απελευθέρωσης των εισαγωγών γεωργικών προϊόντων που προέρχονται από αναπτυσσόμενες χώρες, ε, δυνατότητα απελευθέρωσης των εισαγωγών. Βάσει ποιων κριτηρίων και τι πρέπει να γίνει αυτό και τι ακριβώς εννοείται με αυτό. Ε, σας ευχαριστώ πολύ και πάλι για την εργασία σας. Ε, παρακαλώ. Η κυρία Γκρούνη. Ναι, ε, θα απαντήσω για τη δική μου τροπολογία. Πράγματι θέλω να δοθεί μια ιδιαίτερη προσοχή προς τους νέους, γιατί ακόμα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρώ ότι υπάρχουν πολλοί νέοι που τελειώνουν το σχολείο χωρίς ε, τελικά να μπορούν να ενταχθούν στον κόσμο εργασίας. Ε, και νομίζω ότι θα πρέπει να το εξετάσουμε. Τώρα όσον αφορά αυτά τα στάζια εγώ δεν θεωρώ θα πρέπει να συνδέονται κατά ανάγκη με αμοιβή. Είμαι υπέρ της κατάστασης που επικρατεί στη δική μου χώρα. Δηλαδή να υπάρχει αμοιβή για τα στάζα αυτά όταν υπερβαίνουν τη διάρκεια των δύο ή τριών μηνών. Γιατί ε, έχουν μια ιδιαίτερη αποστολή, ιδιαίτερο χαρακτήρα όταν είναι κάτω από δύο μήνες αυτά έχουν μια αξία για τον μαθητευόμενο, όχι για την επιχείρηση. Και πολύ συχνά οι επιχειρήσει αρνούνται να το κάνουν γιατί λένε ότι δεν έχουν αρκετούς ε, νέους κλπ. Υπάρχουν πάρα πολλές δυσκολίες εκ μέρους των επιχειρήσεων ε, όσον αφορά τα στάζα αυτά και θα πρέπει να είμαστε κάπως προσεκτικοί και να αποτελούν μια αληθινή πρώτη εμπειρία για τους νέους αυτούς και να μπορούν στη συνέχεια να τα αξιοποιούν στην, κατά τη διάρκεια των πανεπιστημιακών του σπουδών, στην εξέλιξη των πανεπιστημιακών του σπουδών κλπ. Τώρα, όσον αφορά την αμοιβή, ε, θεωρώ ότι θα πρέπει να είναι ελάχιστη μια αποζημίωση για την περίοδο αυτή όταν είναι στάζ τα οποία ζητούν μια παρακολούθηση. Ε, νομίζω ότι δεν θα πρέπει να συνδέονται κατά ανάγκη με μια οικονομική ανταμοιβή. Δεν είναι αναγκαίο αυτό. Μπορεί να γίνει υπό κάποιους ώρες. Ευχαριστώ πολύ. Ε, Μιλάμε για την τροπολογία 4 και την 20 ε, συμφωνούμε ότι θα πρέπει να μειωθούν οι ε, ανισότητες, αλλά δεν βλέπω πώς θα μπορούσαμε να βάλουμε κάποιο ανώφλι για το ποια θα είναι το ανώτερο ή το ε, κατώτερο. Και με την πέντε συμφωνώ με την αίσθησή σας, αλλά φυσικά υπάρχουν ορισμένοι που δεν μπορούν να απεργήσουν, όπως οι αστυνομία δυνάμεις, ας πούμε, σε ορισμένα κράτη μέλη. Υπάρχει μια εξαίρεση εκεί και πιστεύω πως υπάρχουν εξαιρέσεις ε, ε εν γέννη. Τροπολογία 20 τώρα. Όσον αφορά την εταιρική ευθύνη, δεν είμαι υπέρ και ποτέ δεν ήμουν υπέρ του να είναι αυτό νομικά δεσμευτικό. Υποστηρίζω τι ελάχιστε προδιαγραφέ, αλλά όχι να είναι νομικά δεσμευτικό. Και αυτά τα είπα μόνο γιατί ο σκιώδης μα είναι σε άλλη επιτροπή αυτή τη στιγμή. Και δίνω και πάλι το λόγο στην Γκαμπριέλ Ζήμερ. Α, συγγνώμη. Με συγχωρείτε. Η Κυρία Στένρικ. Η Φραου δεν μπορούσε σήμερα να είναι παρούσα και μου ζήτησε να διαβάσω τη δήλωσή της. Λέει ότι οι τροπολογίες που έχουν υποβληθεί γενικά είναι θετικές ε, καθότι ενισχύουν τη γνωμοδότηση και αναφέρουν κάποια σημαντικά θέματα όπως είναι η παιδική εργασία, τα δικαιώματα των γυναικών ε, και η κοινωνική εταίρη. Υπάρχουν προβλήματα σε τρία σημεία, τα οποία θα ήθελα σύντομα να αναφέρω. Ε, η τροπολογία 4 προτείνει ε, ανώτατο όριο για τα εισοδήματα, τα οποία η κυρία Ζήπλη βρίσκει προβληματικό. Η ε, θέσπιση ορίου είναι δύσκολη, διότι είναι πολύ δύσκολο να καθοριστεί το ύψος και επίσης αυτό δεν ε, θα ε, ωφελήσει αυτούς που βρίσκονται στην κάτω άκρη της ε, κλίμακας εισόδημάτων. Πιο χρήσιμο θα ήταν να καθοριστεί βασικό μισθό. Η άλλη παρατήρηση είναι για την τροπολογία 12. Δεν ξέρω αν η κυρία Ζήπλη διάβασε την αγγλική ή τη γερμανική εκδοχή. Πιθανότητα το θέμα να είναι μεταφραστικό. Στην τροπολογία 12 αναφέρονται η, ε, η επαγγελματική κατάρτιση, η τεχνολογική εκπαίδευση, όχι όμως η κανονική εκπαίδευση. Ε, είναι απαραίτητο τα παιδιά να λαμβάνουν σωστή εκπαίδευση και θα πρέπει να γίνεται σχετική αναφορά. Η κυρία Σίπλε επίση θεωρεί την τροπολογία 13 όχι πολύ καλή, διότι Ε, γίνεται εδώ πέρα απαρίθμηση διαφόρων ομάδων. Ε, οι νέοι και οι γυναίκες όμως δεν θα πρέπει να θεωρούνται περιθωριοποιημένη ομάδα όπως γίνεται στην τροπολογία. Η κυρία Ζίπελ ε, ελπίζει η Επιτροπή να υιοθετήσει με μεγάλη πλειοψηφία την τροποποιημένη έκθεση για να στείλουμε σαφές μήνυμα προς την Επιτροπή Ανάπτυξης. Αυτό είναι το μήνυμα της κυρίας Ζίπελ. Ευχαριστώ η Κάπριελ Να ευχαριστήσω και πάλι για τις παρεμβάσεις ε, που έγιναν για διευκρίνηση των ε, τροπολογιών ε, καθώς και για τις ερωτήσεις. Κάποιες παρατηρήσεις να κάνω. Πράγματι, κατά την μετάφραση προς τα γερμανικά υπάρχουν ανακρίβειες στο κείμενο, συγκεκριμένα στην τροπολογία 12. Στο αγγλικό κείμενο δεν έχει διαγραφεί τίποτα. Έχει γίνει μόνο η συμπλήρωση ε, για την επαγγελματική κατάρτιση. Ε, δεν έχει διαγραφεί δηλαδή η γενική εκπαίδευση. Και γι' αυτό έκανα πριν την παρατήρηση να βασιστείτε στο αγγλικό κείμενο και σε κάποιες άλλες τροπολογίες ε, υπάρχουν κάποια ερωτηματικά. Ε, σχετικά με τη δημιουργία θέσεων ε, απασχόλησης και η ερώτηση σχετικά με την τροπολογία 25. Το θέμα εδώ είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να είναι ανοιχτή απέναντι στις ε, χώρες να μην δημιουργήσει εμπόδια ε, για την ε, εισαγωγή γεωργικών προϊόντων. χωρίς να πρέπει να προστρέξουμε στις συμφωνίες ελεύθερου εμπορίου, τις οποίες θεωρώ προβληματικές. Θα θέλουμε να βοηθήσουμε τις αναπτυσσόμενες χώρες ε, να ε, επιβιώσουν στην ευρωπαϊκή αγορά. Φυσικά σε κάποιες ε, τροπολογίες υπάρχουν διατυπώσεις όπου συχνά σκέφτομαι ναι τι ακριβώς εννοούμε εδώ. Είναι δύσκολο όμως Ε, σε αυτό το σύντομο κείμενο να αποφύγουμε τελείως τις αντιφάσεις. Ε, αναφερθήκατε στο ανώτατο όριο, αναφερθήκατε στα διαστήματα πρακτικής άσκησης. Είναι δύσκολα τα θέματα αυτά. Δεν ήθελα όμως ε, να απορρίψω τις τροπολογίες αυτές από την αρχή, διότι πιστεύω ότι χρειάζονται διευκρίνηση. Κατά τα άλλα, Συμφωνώ με τις τροπολογίες που έχουν υποβληθεί. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Συγκήτρια. Très bien. Alors, ε, ε, Αύριο θα ψηφίσουμε για την ε, γνωμοδότησή σας και προχωράμε στην ημερησία διάταξη με μια νέα ανταλλαγή απόψεων με μια νέα ακρόαση του Επιτρόπου Λάσλο Άντορ. Σας ευχαριστώ που έρχεστε τακτικά στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων. Έχουμε φορτωμένη μερίσια διαταξή για αυτήν εδώ την ε, επαφή, γιατί σήμερα το πρωί υιοθετήσατε ένα, μέσα στο πλαίσιο της, ε, του προγράμματος εργασίας της Κομισιόν για το 2010, υιοθετήσατε τις κατευθυντήριες γραμμές για την απασχόληση και τα μέλη της Επιτροπής ενδιαφέρονται για να ακούσουν ε, την άποψή σας ε, ταυτόχρονα για το πρόγραμμα εργασίας της Κομισιόν για το 2010, τις κατευθυντήριες γραμμές για την απασχόληση, τα αποτελέσματα του, G, του κοινωνικού G20 και το ηφαίστειο σας ε, απαγόρευσε να είστε πραγματικά παρόν αλλά σίγουρα η πνευματική σας συμβολή θα ήταν σημαντική και επίσης θα θέλαμε να ακούσουμε αυτά όσα έχετε να μας πείτε για τις προπτικές ε, μεταρρύθμισης για τους ευρωπαϊκούς του Κοινωνικού Ταμείου και του Ταμείου Συνοχής. Πριν να σας δώσω το λόγο, θα ήθελα να σας πω ποιο είναι το πνεύμα που επικρατεί εδώ σε σχέση με την υιοθέτηση των κατευθυντηρίων γραμμών περί επασχόλησης, γιατί όπως γνωρίζετε, στην τελευταία συνεδρίαση των ε, Προέδρων των Επιτροπών, ε, εξ ονόματος των συναδέλφων, ζήτησε η υιοθέτηση αυτών των κατευθυντήριων γραμμών να αναβληθεί, ώστε το Ευρωκοινοβούλιο να μπορέσει να εργαστεί υπό καλέ συνθήκε ε, και να ασκήσει το νομοθετικό του έργο, γιατί πρόκειται για ένα κρίσιμο έτο ε, από πολλέ απόψει. Κρίσιμο έτο γιατί η κατάσταση από την άποψη του χρονοδιαγράμματο, ανεξάρτητα από όλη την καλή θέληση του ίδιου του Επιτρόπου, δηλαδή εσά του ιδίου Ε, έχει γνωρίσει πολλές καθυστερήσεις λόγω της έναρξης ισχύω της συνθήκη της Ψαβώνας, λόγω της ε, ε, νέας θητείας της Κομισιόν κτλ. Αλλά αυτό που ανέκαθεν αποτελούσε θέμα μεγάλης ισορροπίας ε, φέτος είναι ακόμα πιο δύσκολο για να διατηρήσουμε, τηρήσουμε μάλλον το αρχικά προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα. Οι κατευθύνες γραμμές όπως γνωρίζετε ε, ανακοινώνονται το, στις 15 Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους και σε αυτή την περίπτωση υιοθετήθηκαν μόλις σήμερα. Πράγμα που δυστυχώς δεν άφησε το Κοινοβούλιο να παρέμβει. Στη διάσκεψη των Προέδρων λοιπόν έχει γίνει ένα τέτοιο διάβημα παρόμοιο, πράγμα που μας επιτρέπει να σκεφτούμε ότι και ο πρόεδρος του και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κ. Μπούζεκ, θα απευθυνόταν στον πρόεδρο της Επιτροπής, ούτως ώστε η υιοθέτηση αυτών των κατευθυντηρίων γραμμών να αναβληθεί για τον Οκτώβριο αφού είναι ούτως ή άλλως πολύ διαστοτικές. Είναι το πρώτο συγκεκριμένο εργαλείο για την εφαρμογή της στρατηγικής 2020. Γι' αυτό και είναι τόσο σημαντικές. Και θέλαμε να μπορέσουμε να, επιβα... να, να επηρεάσουμε τα πράγματα σε συνεργασία με τον εισηγητή μας τον κύριο Όρη. Αυτά ήθελα να σας πω πριν να σας δώσω το λόγο σε μια υπόθεση την οποία γνωρίζετε πλέον πολύ καλά. Έχετε το λόγο κύριε Επίτροπε. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι κύριοι βουλευτές. Είναι πραγματικά τιμή μου και όλα είναι και περισσότερο χαρά μου να έρχομαι στην Επιτροπή και να συζητώ ένα μεγάλο φάσμα θεμάτων που αφορούν την απασχόληση και τις κοινωνικές υποθέσεις. Ε, βλέπετε πως πάντοτε κάτι φρέσκο σας φέρνω. Στην 1η Μαρτίου σας έφερα την στρατηγική ε, για το 2020 που μόλις είχε εγκριθεί από την Επιτροπή τότε και τώρα είναι ακόμα πιο φρέσκες οι νέες ολοκληρωμένες κατευθυντήριες γραμμές που μόλις σήμερα το πρωί συζήτησε και ενέκρινε η Κομισιόν. Είναι κάτι που πραγματικά πιστεύω θα πρέπει να είναι στο επίκεντρο της συζήτησης. Αλλά είμαι έτοιμος να μιλήσω και για άλλα θέματα όπως το 2020 όπως αναφέρθηκε στην εισαγωγή και ίσως και κάποιες άλλες πτυχές της στρατηγική για το 2020 γιατί μεταξύ έχουμε προχωρήσει, έχουμε προοδεύσει και είμαι βεβαίως ότι θα ενδιαφέρεστε για μια ενημέρωση και για αυτό το θέμα. Αλλά να ξεκινήσω με το πρόγραμμα εργασίας της Κομισιόν για το 2010. Το βασικά έγγραφα πολιτικής ε, που υιοθετήθηκαν από τότε που ανέλαβε η νέα Κομισιόν ξεκίνησαν με την ε, στρατηγική για το 2020 και να αντικατοπτρίζουν μια νέα πνοή για τις πολιτικές μας και τώρα όλα αυτά πρέπει να μεταφραστούν σε πράξη. Μέσα στο πλαίσιο της στρατηγικής 2020 στον τίτλο έχουμε μια στρατηγική για συνολική ανάπτυξη και τρεις από τις επτά πρωτοβουλίες και δύο από τους ε, πέντε στόχους για, ε, αφορούν ε, την απασχόληση και τις κοινωνικές υποθέσεις και πιστεύω πως αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο μερίδιο ε, εν γέννη για αυτή τη στρατηγική. Αυτά τα κεφάλαια που εστιάζονται στην απασχόληση και στις κοινωνικές υποθέσεις αντικατοπτρίζονται και στο πρόγραμμα εργασίας ε, της Κομισιόν του 2010. Θα πρέπει να γίνουν ε, δράσεις για τις διάφορες πρωτοβουλίες Φλέξ που σας ανέφερα και που αφορούν τον κοινωνικό τομέα, Youth on the Move, Agenda for News, δεξιότητες και απασχόληση και η Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα για την Ένδια. Για να εφαρμοστούν οι στόχοι αυτών των πρωτοβουλειών θα παρουσιάσουμε τις εξής ε, ανακοινώσεις για το 2010. Ανακοίνωση για την απασχόληση των νέων που θα εκθέτει την πολιτική μας για την αύξηση των ευκαιριών απασχόληση για τους νέους θα προωθήσουμε την κατάρτιση και θα βελτιώσουμε τη μετάβαση από την, παιδεία, από την εκπαίδευση στην εργασία. Αυτή η ανακοίνωση θα, θα, θα, θα παρουσιαστεί σύντομα με την πρωτοβουλία Youth on the Move, νεότητα σε κίνηση από την κυρία Ανδρούλα Βασιλείου. Ε, τα πανεπιστήμια μας καθώς και τα τριτοβάθμια μας εκπαίδευση γενικότερα θα προσελκύσει περισσότερο κόσμο και θα δώσει περισσότερη επασχόληση στους νέους. Επίσης θα παρουσιάσω μια ατζέντα για τις νέες δεξιότητες και, και θέσεις έτσι ώστε να στόχο έχουμε να εξυγχρονίσουμε την αγορά εργασίας, να προωθήσουμε την κινητικότητα και τη διαβίου κατάρτιση και μάθηση. Ε, συμμετοχή στην αγορά εργασίας ε, που θα αντιστοιχεί καλύτερα στην ε, ζήτηση. Αυτό ελπίζουμε πως θα μας βοηθήσει να φτάσουμε το στόχο για την απασχόληση το 2020 που είναι 75% απασχόληση όπως ξέρετε για άνδρες και γυναίκες από τα, για, για τις ηλικίες 20 με 64. Η δεύτερη πρωτοβουλία είναι μια ευρωπαϊκή πλατφόρμα για την καταπολέμηση τη ένδυα. Στόχος είναι να διασφαλίσουμε ότι τα ωφέλη της ανάπτυξης και της ε, ε, ε, ευημερία θα επηρεάζουν όλους. Θα φτάνουν μάλλον σε όλους. Εξάλλου το έτος 2010 είναι το ευρωπαϊκό έτος καταπολέμησης της ένδυας και του κοινωνικού αποκλεισμού. Η ένδυα ε, βρίσκεται σε μεγάλη προτεραιότητα μέσα στο πλαίσιο της στρατηγικής 2020 ώστε να... ο στόχος είναι να βγουν 20 εκατομμύρια άνθρωποι από τη φτώχεια μέχρι το 2020. Όπως γνωρίζετε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έχει ζητήσει να γίνει περισσότερη δουλειά για τους δείκτες, για τους στόχους ε, μείωσης της φτώχειας ε, μέχρι την επόμενή του συνεδρίαση τον Ιούνιο η Κομισιόν συνεργάζεται με τα κράτη-μέλη πολύ εντατικά μέσα στο πλαίσιο της Επιτροπής Κοινωνικής Προστασίας και Κοινωνικής Πρόνοιας αλλά και διμερώς για να διευκρινιστούν όλα αυτά τα θέματα που, όπου περιλαμβάνονται τόσο ευρωπαϊκοί όσο και εθνικοί στόχοι. Η δουλειά προχωρά πολύ και είμαι έτοιμος να απαντήσω σε περαιτέρω ερωτήσει αν το επιθυμείτε γιατί είναι πολύ σημαντική η δουλειά μας εκεί. Το πρόγραμμα εργασία της Κομισιόν επίση τονίζει την δημιουργία μιας ατζέντα των πολιτών, πράγμα που τοποθετεί του ανθρώπου στην καρδιά της ευρωπαϊκής δράσης. Και θα ήθελα να τονίσω τις εξή πρωτοβουλίε. Έχουμε τις προτάσεις για αναθεώρηση τη εργασία για τον χρόνο εργασία, που τη γνωρίζετε καλά, την, ε, επίσης την οδηγία για την απόσπαση των εργαζομένων. Έχουμε διάφορες ε, προ, ε, προκλήσεις μπροστά μας, όπως η γύραση του πληθυσμού. Ένα πράσινο βιβλίο θα δημοσιευθεί τον Ιούνιο για την βιωσιμότητα των συνταξιδοτικών μας συστημάτων. Εστιάζει στην βιωσιμότητα, αλλά και καλύπτει ένα ευρύτερο φάσμα θεμάτων αυτό το πράσινο βιβλίο, γιατί συζητά για τα δημογραφικά θέματα, τη μεταρρύθμιση των συντάξεων και τον αντίκτυπο της ε, χρηματοπιστωτικής κρίσης στις συντάξεις. Ως μη στρατηγική πρωτοβουλία να σας ε, θυμίσω επίσης ε, το θέμα της έκθεσης στη ηλεκτρομαγνητικά πεδία. Επίσης τέτοια οδηγία θα συζητηθεί στην ατζέντα υγείας και ασφάλειας Πρέπει να βρεθεί μια λύση επιγόντω. αν θέλουμε να, να διευκρινίσουμε την νομική κατάσταση σε διάφορα κράτη-μέλη, γιατί όπω γνωρίζετε έχω ξεκινήσει την πρώτη φάση διαβούλευση με του κοινωνικού εταίρους και προσβλέπω στη συμβολή του ώστε να μπορέσουμε να προχωρήσουμε με αυτή τη συζήτηση επικοδομητικά. Όσον αφορά την οδηγία για την απόσπαση των εργαζομένων, η Κομισιόν αυτή τη στιγμή εξετάζει τι διάφορε επιλογέ για την αντιμετώπιση των δυσκολιών εφαρμογή συμπεριλαμβανομένων κάποιων από αυτούς που προκύπτουν λόγω των, τρίτων, των υπηκών τρίτων χωρών. Θα πρέπει ε, όλα αυτά να μας απασχολήσουν μέχρι το 2011. Όσον αφορά τώρα τον κανονισμό, την, την ατζέντα για την έξυπνη, ε, ε, ε, έξυπνους κανονισμούς, θα επιταχύνουμε την εργασία μας, ώστε να, αλλά και τον έλεγχό μας όσον αφορά, για, για, να δούμε την αποτελεσματικότητα των πολιτικών μας. Ένα άλλο θέμα στο πρόγραμμα εργασίας είναι το μέλλον του προϋπολογισμού της Ένωσης. Η αναθεώρηση της, ε, του προϋπολογισμού θα μας δείξει πώς το νέο δημοσιονομικό πλαίσιο θα μπορούσε να συμβάλλει στις προτεραιότητες 2020. Θα μεριμνήσω ώστε να οδηγηθούμε σε ένα νέο ε, σχηρότερο κοινωνικό ταμείο που θα εστιάζει στον, στους ανθρώπους και στην απασχόληση. Θέλουμε οι άνθρωποι να μπορούν να ξεκινήσουν την εργασία, να παραμείνουν απασχολούμενοι. Ε, μιλάμε για 10 εκατομμύρια, ε, πολλά εκατομμύρια ευρώ ετησίω και βοηθάμε με αυτό το πρόγραμμα 10 εκατομμύρια ανθρώπου ετησίω να βελτιώσουν την κατάστασή τους. Παρά την κρίση, τα κράτη-μέλη τα έχουν πάει σχετικά καλά ε, όσον αφορά τι πολιτικέ απασχόλησης και την διαβίου κατάρτιση. Η Κομισιόν συμβάλλει ενεργά ε, και βοηθά αυτές τις χώρες που υστερούν. Ε, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο έχει αποδείξει την αξία του σε αυτή την ε, κρίση. Έχουμε βελτιώσει την πρόσβαση στο Ταμείο, βελτιώσει την πρόσβαση στο Ταμείο και το έχουμε καταστήσει πιο αποτελεσματικό. Επίσης έχουμε απλοποιήσει τις διαδικασίες μας ώστε τα χρήματα να δίνονται, τα κονδύλια να δίνονται πιο εύκολα και έχουμε φτιάξει ε, και τη δυνατότητα ε, δανεισμού για 100 εκατομμύρια ευρώ έτσι ώστε να μπορούν διάφοροι να βρουν ευκολότερα λύση και να βγουν από την φτώχεια. Μάλιστα, εχθές συζητήσαμε πιο ε, λεπτομεριακά πώς θα μπει στη λειτουργική της φάση αυτή η δυνατότητα για μικροδάνεια. Τώρα, για τις ολοκληρωμένες κατευθυντήριες γραμμές, κυρία Πρόεδρε, σήμερα ε, ε, υιοθετήθηκαν είναι ένα σύνολο 10 κατευθυντήριων γραμμών, 4 εκ των οποίων στον τομέα της απασχόλησης και των κοινωνικών υποθέσεων με στόχο περισσότερες και καλύτερες θέσεις απασχόλησης και συμβολή στην έλλειψη αποκλεισμού. Είναι ένα ισορροπημένο πακέτο που η απασχόληση και τα κοινωνικά ζητήματα έχουν μεγάλο βάρος. Οι προτινόμενες κατευθυντήριες γραμμές έχουν στόχο να αυξήσουν τη συμμετοχή στην αγορά εργασίας, να μειώσουν τη διαστατική ανεργία μέσω ολοκληρωμένων και ισορροπημένων πολιτικών ευελιξίας. Επίσης, στόχο έχουν να αναπτύξουν ένα εργατικό δυναμικό με πολλές δυνατότητες ώστε να, ε, να αντιστοιχούν οι εργαζόμενοι στη ζήτηση της αγοράς. Μια από τις καινοτομίες είναι η συμπερίληψη μιας κοινωνικής κατευθυντήρες γραμμής με τη στόχο την καταπολέμηση της στόχιας και το κοινωνικού αποκλεισμού μέσω της πρόσβασης σε υπηρεσίες υψηλής ε, ποιότητας, Καθώ και τον εξυγχρονισμό των ε, συστημάτων κοινωνική ασφάλιση και συνταξιοδότηση. Η συμβολή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι ζωτική σημασία. Πρέπει να ληφθεί υπόψη, πράγμα που σημαίνει ότι το Κοινοβούλιο χρειάζεται χρόνο για να συντάξει μια γνωμοδότηση. Για να έχει το Κοινοβούλιο αρκετό χρόνο, η τελική αξιολόγηση, επικύρωση μάλλον τη στρατηγική, θα υποβληθεί στο Συμβούλιο μετά από τι καλοκαιρινέ διακοπέ. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα εγκρίνει μόνο από πολιτική πλευρά τι κατευθυντήριες γραμμέ και θα αυτές θα εγκριθούν επισήμως από το Συμβούλιο μόνο όταν θα έχουν ληφθεί η γνωμοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου επί των ε, κατευθυντηρίων γραμμών περί επασχόλησης. Ένα άλλο σημείο που θέλω να καλύψω είναι το αποτέλεσμα της ε, ε, συνεδρίασης των Υπουργών στην Washington, πράγμα που ανέφερε η Πρόεδρος, όπως σας είπα, δυστυχώς Ήμουν ο πρώτος Ούγγρος πολιτικός που δεν κατάφερε να πάει στο G20 λόγω του ηφαιστείου. Ωστόσο θεωρούμε πολύ θετικό το γεγονός ότι συνεδρίασαν οι Υπουργοί Απασχόλησης με την εξαίρεση κάποιων Ευρωπαίων, ήταν ο Γερμανός, ο Βρετανός, εγώ, επικεφαλής του ΩΣΑ και διάφοροι άλλοι. Εν πάση περιπτώσει ήταν μια πολύ σημαντική κίνηση γιατί αυτή η υπουργική διάσκεψη εξέτασε πολιτικές και μέτρα στον τομέα της απασχόλησης και των κοινωνικών πολιτικών και στόχο είχε να βελτιώσει την ποσότητα αλλά και την ποιότητα των θέσεων απασχόλησης και το πώ θα προετοιμαστούμε για την οικονομία μετά την κρίση. Προέκυψαν ε, πολύ στεναρές συστάσεις, καλύπτουν την ανάγκη να επιταχυνθεί η δημιουργία θέσεων απασχόλησης, να τεθεί στο επίκεντρο των εθνικών και παγκόσμιων οικονομικών στρατηγικών η εξάλληψη της στόχη και του κοινωνικού αποκλεισμού. Επίσης τονίζεται η ανάγκη να βελτιωθούν, να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις μέσω προτεραιότητας στην παιδεία, τη διαβίου κατάρτιση και την ε, συμμετοχή καθώς και την αντιστοιχεία δεξιοτήτων και θέσεων απασχόλησης. Γενικώ ε, θα έχουν γίνει προτάσεις για τη βιώσιμη και μόνιμη ανάπτυξη. Θα υποβληθούν στο Τορόντο το καλοκαίρι όλα αυτά και νομίζω πως μπορούμε να είμαστε ικανοποιημένοι για τον τρόπο με τον οποίο ε, έγινε δεκτή η συμβολή μας, η οποία μεταφέρει τις ευρωπαϊκές αξίες. Κυρίε και κύριοι, είναι πρόθεσή μου να εξακολουθήσω να έρχομαι στο σώμα για τα θέματα όλα αυτά, της απασχόλησης και, των, ε, κοινωνικό, και κοινωνικής πρόνοιας. Έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας, αν θέλουμε να πετύχουμε την κοινωνία που επιθυμούμε και που έχουμε περιγράψει μέσα στη στρατηγική 2020. Οι ουρανοί της Ευρώπης είναι συνεφιασμένοι λόγω πολλών ε, προκλήσεων. Και αυτό δεν σημαίνει μόνο ε, ε, ε, τη στάχτη από το ηφαίστειο, αλλά και την οικονομική και χρηματοπιστωτική σταθερότητα, η οποία δεν είναι πάντα δεδομένη. Πρέπει να καταβάλουμε πολύ περισσότερες προσπάθειες για να την επιτύχουμε, να έχουμε σταθερότητα, να έχουμε οικονομική ανάκαμψη να δημιουργήσουμε εκ νέου θέσει στην επόμενη περίοδο. Πιστεύω πως το πρόγραμμα εργασίας το οποίο σας περιέγραψα είναι σχεδιασμένο για να ε, αντιμετωπίσει αυτές τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε στο δικό μου το χαρτοφυλάκιο και έχουμε στόχο να συνεργαστούμε στενά με το Κοινοβούλιο στην εφαρμογή αυτών των κατευθυντηρίων γραμμών. Σας ευχαριστώ πολύ και είμαι έτοιμος να απαντήσω σε ερωτήσεις σας. Ευχαριστούμε πολύ αγαπητά κύριε Πίτροπε. Υπάρχουν 21 συνάδελφοι που θέλουν να πάρουν το λόγο. Δεν ξέρω ποιος δεν ζήτησε να πάρει το λόγο. Θα σας ε, προτείνω για να μπορεί ο καθένας να πάρει το λόγο να πάρουμε ομάδες τεσσάρων ερωτήσεων. Θα δώσω καταρχήν το λόγο στους συντονιστές των ομάδων που μου τον ζήτησαν, αλλά πριν το κάνω θα ήθελα να επωφεληθώ τις θέσεις μου της, ως Προέδρου για να κάνω καταρχήν μια παρατήρηση και να σας θέσω ένα ερώτημα. Η παρατήρηση έχει ως εξή. Κατανοώ τα όσα μας είπατε, δηλαδή ότι επιθυμείτε ότι ε, οι κατευθυντήριες για την απασχόληση ε, θα εγκριθούν το φθινόπερο. Αλλά είπατε ότι η πολιτική συμφωνία θα μπορούσε ήδη να επιτευχθεί τον Ιούνιο. Και για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τι σημαίνει κάτι τέτοιο, τι σημαίνει πολιτική συμφωνία. Πολιτική συμφωνία είναι όσα αποφασίζει το Συμβούλιο χωρίς να ακούσει το Κοινοβούλιο. Νομίζω ότι τα πράγματα δεν πάνε έτσι ε, καλά και είμαστε διατεθειμένοι να συνεργαστούμε με τις βαλικές αρχές που θα έχουν την ευθύνη πριν ε, από το Συμβούλιο του Φθινοπόρου. Και αυτό είναι ένα θέμα ιδιαίτερο σημαντικό για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Εάν δεν ληφθούν υπόψη οι θέσεις του Κοινοβουλίου από το Συμβούλιο, θεωρούμε ότι δεν έχει προηγηθεί κανένας διάλογος και θα αντλήσουμε τις νομικές ε, συνέπειες και νομίζω ότι επί τούτου υπάρχει μια πλατεία συνένεση των πολιτικών ομάδων. Έστω και αν κατανοούμε ότι βεβαίως ε, θα υπάρξει ένα συμβούλιο το φθινόπωρο ε, αλλά ε, υπάρχει μια πολιτική συζήτηση αλλά δεν είναι δυνατόν να πάψει, να σταματήσει η πολιτική συζήτηση εάν δεν έχει ζητηθεί και η γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Το ερώτημά μου αφορά τις εκθέσεις αξιολόγησης που κάνατε με τους με συναδέλφους στο Επίτροπο Περιφερειακής Ανάπτυξης όσον αφορά τον απολογισμό για το Ταμείο Συνοχής. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό για τα μέλη αυτής της Επιτροπής να μπορέσετε να μας κάνετε έναν απολογισμό γιατί όλοι υπερασπιζόμαστε αυτό το θέμα, ωστόσο η ένταξή μας σε μια σφαιρική οικονομική στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης πραγματικά έχει πολλές ελλείψεις και η λειτουργία της ε, δεν μας επέτρεψε μέχρι στιγμής να βοηθήσουμε τις χώρες που είχαν ανάγκη πριν από την κρίση και που όπως φαίνεται τελικά ε, πυροδοτήθηκε από την ίδια την κρίση. Θα θέλαμε να είχαμε την άποψή σας για αυτό το θέμα. Θα δώσω το λόγο λοιπόν στους συντονιστές, καταρχήν στον κύριο Ρή. Θα τους αφήσω να μιλήσουν λίγο παραπάνω και στη συνέχεια βεβαίως θα, κάνουμε την, θα έχουμε τη συζήτηση. Ε, και... Πρόεδρε, θα ήθελα να καλωσορίσω και εγώ τον Επίτροπο. Είπατε, Πρόεδρε, αυτό που ήθελα να πω και εγώ, συμφωνώ απόλυτα με τη θέση που περιγράψατε. Είχαμε μεγάλη συζήτηση εντός του ΕΛΚ και ήταν σαφής η θέση ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι διατεθειμένο να προχωρήσει όσο μπορεί σε περίπτωση που μας αγνοήσουν τόσο πολύ όσο είδαμε και εάν δεν ε, γίνεται σεβαστός ο κανονισμός του Κοινοβουλίου. Δεν μιλάμε για ανικανότητα εκπόνησης νομοδοτήσεων του Κοινοβουλίου. Το Κοινοβούλιο μπορεί μόνο να διαμορφώσει θέση εάν οι βουλευτές έχουν το χρόνο να συζητήσουν τα θέματα, να τροποποιήσουν τα κείμενα και να τα ψηφίσουν. Είναι μια διαδικασία που απαιτεί κάποιο χρόνο. Η πρόσφατη διαδικασία δεν μας επέτρεψε να ακολουθήσουμε τον κανόνα αυτό. Η θέση μας λοιπόν ευθυγραμμίζεται απόλυτα με τη δήλωσή σας, κυρία Πρόεδρε. Είναι πολύ σωστά αυτά που ακούσαμε. Συμφωνούμε ότι τα θέματα που θύχτηκαν είναι πολύ σημαντικά. Η συμμετοχή νέων και ηλικιωμένων, η ένταξή τους στην απασχόληση είναι σημαντική. Δεν συμφωνούμε απόλυτα με τη θέση σας όσον αφορά την οδηγία για τις αποσπάσεις, για τους αποσπασμένους εργαζομένους. Επικροτούμε γι' αυτό την πρόσφατη δήλωση της Επιτροπής ότι μπορεί να τροποποιηθούν οι κανόνες και το ΕΛΚ θα υποστηρίξει την προσέγγιση αυτή. Νομίζω ότι είναι σημαντικό να επανεξεταστούν ε, τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία, διότι η τεχνολογία αλλάζει γρήγορα και θα πρέπει να αντιδρούμε, να αναθεωρούμε δηλαδή και να προσαρμόζουμε τους κανόνες μας ανάλογα. Όσον αφορά την πράσινη βίβλο για την βιωσιμότητα των συντάξεων, έχουμε μεγάλες προσδοκίες. Είμαι βέβαιος ότι θα γίνει μεγάλη συζήτηση, είναι θέμα κλειδί και το ΕΛΚ θα ε, συμβάλλει επικοδομητικά στη συζήτηση αυτή. Έχω κάποιες ερωτήσεις. Μέχρι τώρα δεν έχουμε συζητήσει τη χρηματοδότηση. Στην συζήτηση για τη στρατηγική 2020 ε, βλέπουμε κάποια δύναμα σημεία όσον αφορά το, την απασχόληση επειδή δεν έχουμε ακούσει τίποτα σχετικά με τη χρηματοδότηση. Το μόνο που ξέρουμε είναι ότι η χρηματοδότηση θα πρέπει να είναι προσαρμοσμένη στη στρατηγική, αλλά δηλαδή δεν έχουμε λεπτομέρειε σχετικά με το πώ θα γίνει αυτό. Όσον αφορά τι δηλώσει του Επιτρόπου, μπορώ να συμφωνήσω απόλυτα. Στο ΕΛΚ είχαμε συζητήσει για το θέμα αυτό και συμφωνήσαμε ότι η πολιτική συνοχή θα πρέπει να έχει ειδικό βάρος στα πλαίσια της στρατηγικής του 2020 και ιδιαίτερα ε, στο τομέα της απασχόλησης. Θα πρέπει να επανεξεταστούν λοιπόν τα κοινωνικά ταμεία, θα πρέπει να συμπεριληφθούν στο πακέτο του προγράμματος. Μπορείτε λοιπόν να βασιστείτε στην υποστήριξή μας. Να είσαστε βέβαιος ότι θα σας υποστηρίξουμε. Ένα άλλο θέμα είναι η έλεγχη και τα αντίβαρα, διότι στα πλαίσια της στρατηγικής της Λισαβόνας έχουμε κατευθυντήρες γραμμές. Τα κράτη-μέλη έχουν ε, ε, υποβάλει αναφορές σχετικά με την εφαρμογή των κατευθυντηρίων γραμμών. Ε, το αποτέλεσμα δεν είναι τελείως αποκαρδιωτικό. Δεν συμφωνώ με αυτούς που λένε ότι δεν υπάρχουν καθόλου αποτελέσματα, διότι υπήρχαν κάποια θετικά αποτελέσματα τα οποία βέβαια αντιστάθμισε η κρίση. Θα πρέπει να εξετάζουμε την εκπλήρωση των στόχων μας και θα ήθελα να επικροτήσω το γεγονός ότι ε, θέλετε να συγκεντρώσετε την προσοχή μας στην αναθεώρηση των φορολογικών προγραμμάτων, διότι αν θέλουμε να δημιουργήσουμε μεγάλο αριθμό νέων θέσεων απασχόλησης, ε, τα φορολογικά καθεστώτα θα πρέπει να προσαρμοστούν ανάλογα. Πιστεύω ότι η Κομισιόν θα πρέπει να το προσέξει αυτό. Ευχαριστώ. Ο κύριος Σέρκας και στη συνέχεια η κυρία Λίν, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θα είμαι πιο σύντομος από συνάδελφα, αλλά ωστόσο θα υπάρξουν πολλοί σοσιαλιστές συνάδελφοι που θα συμπληρώσουν τα όσα λέω εγώ. Καταρχήν, κύριε Επίτροπε, καλώ ήρθατε στην Επιτροπή μα και πάλι και θα ήθελα να σα ευχαριστήσω ειλικρινά για όλη την προσπάθεια που καταβάλλετε για να τοποθετήσετε τα ζητήματα απασχόληση και τα κοινωνικά ε, θέματα στο επίκεντρο τη ε, προσοχή τη Επιτροπή. Ε, και οι ευχαριστίε μου λοιπόν σχετίζονται βεβαίως, συνοδεύονται από την κατανόηση ότι το έργο σας είναι εξαιρετικά δύσκολο. Γιατί σήμερα ε, λέγονται πολλά για τα ζητήματα απασχόλησης. Ε, δεν βρίσκονται δυστυχώ στο επίκεντρο της προσοχής της Ευρώπης. Ε, εμείς παρόλα αυτά ε, βλέπουμε ότι έχουν γίνει κάποιες ε, πρόοδοι έχει γίνει ένα βήμα προς τα μπρος, ειδικά με τη συνάντηση της Washington και ε, δεν ήταν μόνο μια συνάντηση ηγετών, ε, φίλων ή συναδέλφων, αλλά θα πρέπει η συνάντηση αυτή να περάσει, να εφαρμοστεί και στην πραγματικότητα, ούτω ώστε, η πραγματική εξωτερικο... το κοινωνικό μοντέλο όντως να μειώσει την ε, φτώχεια. Αυτή είναι μια πραγματικότητα την οποία ζητούμε από την Επιτροπή να ασκήσουμε μια πίεση προς αυτή την κατεύθυνση ωστόσο δεν συμπεριλαμβάνεται κάτι τέτοιο στο πρόγραμμα της Επιτροπής. Λέγονται πολλά, αλλά όταν πρέπει να γίνει το πέρασμα στην πράξη υπάρχει μια τεράστια απόκληση από τις θεωρίες στην πράξη. Και ε, γιατί το Συμβούλιο και η Επιτροπή ακόμα δεν καταλαβαίνουν, δεν κατανοούν ότι η κρίση από την οποία υποφέρει η Ευρώπη, η κρίση από την οποία πάσει ο κόσμος απαιτεί μια, έναν τεράστιο ε, συμβιβασμό όχι μόνο ρητορική ε, φύσεως αλλά ένα πέρασμα στην πράξη. Θα πρέπει να ληφθούν κάποιες επώδυνες αποφάσεις. Ε, σήμερα βλέπουμε την κρίση από την οποία υποφέρει η Ελλάδα και την κρίση στην αγορά απασχόληση σε πάρα πολλές χώρες. Κύριε Επίτροπη, εκτός από εσά, ποιοι επίτροποι πιστεύουν ότι είναι πιο σημαντικό να λυθούν τα προβλήματα αυτά πραχυπρόθεσμα και να μην ε, περιμένουμε η ίδια η αγορά εργασίας να επιλύσει τα τεράστια προβλήματα εκατομμυρίων εργατών που έχασαν τη θέση απασχόλησης. Ε, ε, κλείνω κυρία Πρόεδρε. θα ήθελα να σας θέσω ένα ερώτημα σε σχέση με δύο θέματα θεμελιώδη. Η οδηγία της των αποσπασμένων εργαζόμενων και του χρόνου εργασίας. Γιατί είναι οι πολίτες οι οποίοι βρίσκονται, ε, τους αφορά αυτή η οδηγία. Και οι λύσεις που δίνει αυτό το κοινοβούλιο τελικά θέτουν τους εργαζόμενους στο επίκεντρο. Νομίζω ότι θα πρέπει να υπάρξει μια συμφωνία μεταξύ Επιτροπής και Συμβουλίου εν σχέση με τις πολύ σημαντικές αυτές ε, οδηγίες. Ευχαριστώ. Κυρία ε, Λίν, ε, πράγματι η οδηγία για τις αποσπάσεις των γαζομένων ε, θέτει το ερώτημα κατά πόσο χρειαζόμαστε περισσότερε κατευθυντήριες γραμμέ ή ε, ε, ανάγκη εφαρμογή. Τώρα, όσον αφορά τις συντάξεις, θα ήθελα να δω να γίνονται κάποια πράγματα μακροπρόθεσμα. Τώρα, η οδηγία για τα μαγνητικά πεδία. εργάστηκα πάρα πολύ με τον Επίτροπο κ. Σπίτλερ, συνεργάστηκα και τα προηγούμενα χρόνια και ήταν σαφές ότι θα πρέπει να υπάρξει ένα μορατόριο. Ε, και θα ήταν ενδιαφέρον να μας πείτε κι εσείς τι προτίθεστε να κάνετε και κατά πόσο θα υπάρξουν αυτά τα σκάνες ε, υγείας ε, σε σχέση με την, τα MRI scanners τα οποία καλύπτονται από την οδηγία για τις ιατρικές συσκευές. Ξέρω ότι υπάρχουν κάποια προβλήματα. Δεν ξέρω τι θα γίνει με την οδηγία για τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία. Θα υπάρξει μια οδηγία η οποία εξαγγέλθηκε ε, το Μάιο από την Επιτροπή um, για τα μειοσκελετικά προβλήματα. Και ε, διερωτώ ε, τι θα γίνει με αυτή την οδηγία που ακριβώς ε, βρισκόμαστε. Καθώς υπάρχουν πολλά ερωτήματα, θα ήθελα κύριε Επίτροπε να απαντήσετε πραγματικά εν συντομία, αλλά βεβαίως να καλύψετε όλες τις ερωτήσεις. Ναι, ε, μια ερώτηση Συνοχή είναι πολύ δύσκολο να απαντηθεί με έναν ε, επιγραμματικό τρόπο. Παρ' όλα αυτά θα ήθελα να τονίσω ότι είναι ένα θέμα, μια πολιτική θεμελιώδη σημασία που αφορά ένα θεμελιώδη εργαλείο, ένα θεμελιώδη μηχανισμό για την Ευρωπαϊκή Ένωση και ε, δεν θα πρέπει να γίνει σπεσμένα η κρίση και αξιολόγηση. Θα πρέπει να δούμε πώς στις ε, χώρες του Ταμείου Συνοχής τα ταμεία συνοχής και τα διαρθρωτικά ταμεία ε, παίζουν ένα, μπορούν να διαμερίσουν ένα ζωτικό ρόλο όσον αφορά την ενίσχυση των επενδύσεων και την αναζωγόνηση του επιχειρηματικού πνεύματος και την υποστήριξη ε, των υποδομών, χωρίς οποίες είναι αδύνατο να υπάρξει ανάπτυξη. Έστω και μικρής κλίμακα ανάπτυξη των υποδομών ε, μπορεί να είναι εξαιρετικά δυσχερής χωρίς τα κονδύλια που παρέχει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι λοιπόν ε, πιστεύω και συμφωνώ εδώ με τον ε, Μόδιο Επίτροπο. Θα πρέπει να έχουμε κατά πάσα πιθανότητα εξελογή σε πιο τακτική βάση. Θα πρέπει να ενισχύσουμε το κύκλο των αξιολογήσεων, ούτε ώστε να έχουμε ένα ταχύτερο, γρηγορότερο feedback προς αυτούς που εκπονούν τα προγράμματα και συγκεντρώνουν τις εμπειρίες από τις χώρες που αξιοποιούν αυτά τα κονδύλια, τα ταμεία. Αλλά από την άλλη θα πρέπει να υπάρχει μια σαφήνεια χωρίς αμφισημίες, χωρίς ε, ε, σκοτεινά σημεία, γιατί είναι βασικός πυλώνας της ε, πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. τώρα, ας συνεχίσουμε με ζητήματα χρηματοδότησης και χρηματοπιστωτικού εργαλείου. Σήμερα ο Επίτροπος κ. Λεβαντόφσκι αναφέρθηκε σχετικά στο πλαίσιο του επόμενου προϋπολογισμού και είναι απολύτως ξεκάθαρο ότι οι προτάσεις για τον προϋπολογισμό συνδέουν το χρηματοπιστωτικό εργαλείο με τις ευέλικτες ε, πρωτοβουλίες που θα υπάρξουν μελλοντικά σε σχέση ακριβώς με αυτή την χρηματοδοτική δυνατότητα αλλά θα πρέπει να εξασφαλίσουμε οι πρωτοβουλίες αυτές στον κοινωνικό τομέα να έχουν επαρκή χρηματοδότηση μέσω του κοινωνικού ταμείου. Αυτό είναι κάτι το οποίο λαμβάνουμε υπόψη ακριβώς στο πλαίσιο της ε, αναθεώρησης του προπολογισμού που αποτελεί έργο των προσεχών μηνών. για τον κύριο Σέρκα θα ήθελα να πω ότι είναι πολύ δύσκολο να απαντηθεί το ερώτημά του επιγραμματικά. Οι πυλώνες της Ευρώπης 2020 και αυτό ε, είναι ένα θέμα που, στο οποίο συμφωνούν όλοι οι επίτροποι, όλοι υποστηρίζουμε μία ατζέντα η οποία δεν ε, θέλει μόνο μια βιώσιμη ανάπτυξη, αλλά μια ανάπτυξη που αναλαμβάνει και την κοινωνική πτυχή, την κοινωνική ανάπτυξη της Ευρώπης. Και αυτό εκφράζεται, για παράδειγμα, όχι μόνο σε στήματα πολιτικής απασχόλησης και κοινωνικής πολιτικής, αλλά επίσης έχουμε μπροστά μας ε, τα ζητήματα των ε, οικονομικών κανονισμών. Ο Επίτροπος ε, κ. Μπαρνέα ασχολείται με τα θέματα αυτά της ε, χρηματοπιστωτικής σταθερότητας που θα απαλείψει την υπάρχουσα βεβαιότητα στον ευρωπαϊκό χώρο και θα επιτρέψει ένα νέο μια νέα κατάσταση. Χωρίς τη δημιουργία χρηματοπιστωτικής ε, σταθερότητας δεν είναι δυνατόν να υπάρχουν νέες επενδύσεις και δεν θα έχουμε μια στέρεη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Αυτός είναι ένας τομέας ε, όπου δεν απόκειται μόνο στην αρμοδιότητά, του, αρμοδιότητά μου αλλά εμπίπτει στη συντονισμένη αρμοδιότητα πολλών γενικών διευθύνσεων. Ε, αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε μια κρίσιμη φάση όσον αφορά τον διάλογο με τους κοινωνικούς εταίρους ε, και θα δω τους ηγέτες των επιχειρηματικών κύκλων για να συζητήσουμε ε, ορισμένα από αυτά τα θέματα και θα κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου για να συμπεριθούν και απόψεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και αν δεν γίνει αυτό δεν θα γίνουν τα επόμενα βήματα. Παρ' όλα αυτά θα πρέπει να γίνουν κάποια βήματα γιατί δόθηκε η υπόσχεση από τον ε, Πρόεδρο. Όσον αφορά το G20, η Επιτροπή ενθαρρύνει τις χώρες μέλη να επικαιρώσουν ε, τη σύμβαση της ILO και αυτό κατά την άποψή μας είναι κάτι το οποίο ε, γίνεται σε επίπεδο, θα να γίνει σε επίπεδο χωρών μελών και παρακολουθούμε εκ του σύνεγγυς τις εξελίξεις στο επίπεδο των ε, χωρών μελών και προσπαθούμε να τις ενθαρρύνουμε. Όσον αφορά τα άλλα θέματα, ε, σε σχέση με τα νομοθετικά θέματα στο χώρο υγιεινής και ασφάλειας, στην ημερήσια διάταξη αυτού του έτους έχουμε το θέμα της έκθεσης στην ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία και δυστυχώς έχουμε αναβάλει για το επόμενο έτος την πρωτοβουλία για τις μυοσκελετικές διαταραχές αλλά θα αποτελέσει μία από τις στρατηγικές πρωτοβουλίες του επόμενου έτους. Θα πρέπει λοιπόν να εντοπίσουμε, να κάνουμε τη διάκριση μεταξύ των στρατηγικών θεμάτων αυτού του έτου και του επόμενου. Αυτό το έτος είναι η καταπολέμηση της φτώχειας και η δημιουργία νέων δεξιοτήτων και για το επόμενο έτος έχουμε τις προτάσεις για τις μυοσκελετικές διαταραχές ε, που θα μας απασχολήσουν στις αρχές του επόμενου χρόνου. Ευχαριστώ. Θα ακούσουμε δύο συντονιστές, την κυρία Λαμπέρ και την κυρία Τσίμερ στη συνέχεια. Ευχαριστώ Πρόεδρε και ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Νομίζω ότι αυτό που υπονοήθηκε είναι ότι θα δούμε αρκετές εντάσεις στις κατευθυντήρες γραμμές. Ε, ανάμεσα στην πτυχή της απασχόλησης και στην οικονομική. Ε, πόσο μάλλον για τα θέματα ε, ελλείμματος στον προϋπολογισμό και πώς θα ταιριάξει αυτό με την ανάγκη για ισχυρές δημόσιες υπηρεσίες και πώς ταιριάζει αυτό με το σχέδιο του Συμβουλίου για την ενεργό ένταξη. Πώς θα φροντίσουμε να μην υποφέρουν οι δημόσιες υπηρεσίες λόγω της επίδρασής τους στην ατζέντα κατά της ένδυας. Όσον αφορά τη στρατηγική του 2020, μου φαίνεται ότι έχουμε φτάσει σε ένα σημείο όπου μιλάμε για την ανάπτυξη ως αποτέλεσμα και όχι ως μηχανισμό. Ποιοι θα είναι οι δείκτες για θέματα όπως είναι η βιωσιμότητα, διότι εδώ και αρκετό καιρό έχουμε ένα δίλημα ανάμεσα στην δημιουργία θέσεων απασχόλησης και στην ανάπτυξη. Αυτά τα δύο δεν ε, ε, ε, πάνε απαραίτητα μαζί. Έχουμε το θέμα της αύξησης της απασχόλησης. Χαίρομαι που βλέπω ότι μιλάμε για αύξηση της πράσινης απασχόλησης, τη φροντίδα και την πρόθεση της καινοτομίας. Και ελπίζω ότι αυτό θα ταιριάξει με την νέα ε, ατζέντα για τις δεξιότητες, ε, τα επαγγελματικά προσόντα και την κατευθυντήρια γραμμή 4 που αναφέρεται και στη μείωση των εκπομπών. Και μιλάτε επίσης για ένα ισχυρό Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Μπορείτε να μου εξηγήσετε τι εννοείτε με αυτό και ποιο θα φροντίσει να είναι ισχυρό το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, διότι υπάρχουν ανησυχίες ότι υπάρχει αυξανόμενη πανεθνικοποίηση και ότι η προσοχή των ε, κρατών μελών ε, στρέφεται μακριά από αυτό ε, όσο αποκτούν μεγαλύτερο έλεγχο των χρημάτων χωρίς να ενδιαφέρονται για τον για τον έλεγχο των χρημάτων αυτών. Ευχαριστώ κυρία Τσίμερ και κατόπιν ο Τόμας Μαν. Θα ήθελα να συμφωνήσω με την προλαλή σας. Ε, συμμερίζομαι απόλυτα το προβληματισμό της και θα ήθελα να τον αναπτύξω όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Έτος κατά της Ένδυας. Είναι μία εκστρατεία για να πάψει να είναι ταμπού η Ένδυα. Αυτό σημαίνει δηλαδή ότι μέσα στα πλαίσια της κοινωνίας μας θα πρέπει να συνηθίσουμε ότι υπάρχει ένδυα και ότι και θα, πρέπει να υπάρχουν μέτρα για την εκρίζωση της ένδυας. Με ενδιαφέρει λοιπόν τι προετοιμασία, τι εκπαίδευση σχεδιάζει η Κομισιόν ώστε στη διάσκεψη κορυφής του Ιουνίου να οδηγήσει τους ε, αρχηγούς των κυβερνήσεων ε, να ε, ακολουθήσουν τα αποτελέσματα της ε, Συνόδου Κορυφής της Κομεχάγης του 1995 και να αναπτύξουν μια στρατηγική κατά της ένδυας. Θυμάμαι από το, την Σύνοδο, από το Ανοιξιάτικο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο η, ε, η καγκελάριος Μέρκελ είπε ότι είναι κατά οποιασδήποτε θέσπιση στόχου για την ένδυα στην στρατηγική 2020 επειδή η ένδυα είναι θέμα κοινωνικό και έτσι εθνικό. Αυτό πιστεύω ότι είναι σημαντική οπισθοχώρηση. Και όταν κοιτάω αυτά που συμφωνήθηκαν το 1995, πώς θα πετύχουμε να κινητοποιήσουμε τους αρχηγούς των κυβερνήσεων μέχρι την, ε, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του ε, Ιουνίου. Βλέπουμε τις ανακοινώσεις ε, της βελγικής κυβέρνησης, τους στόχους που έχουν θέσει για την ανάληψη της Προεδρίας από αυτούς όσον αφορά την ένδια αναφέρονται στην στήριξη για την κατανάλωση ενέργειας την επιδότηση. Ε, αυτές λοιπόν τις συγκεκριμένε ανακοινώσεις της βελγικής κυβέρνησης ε, πώς ε, μπορούμε να τις δούμε και μαζί με αυτά που λέει η Κομισιόν και με βάση συγκεκριμένους δείκτες και με βάση συγκεκριμένα μέτρα. Ευχαριστώ. Ωραία λοιπόν, τώρα θα περάσουμε στους ομιλητές εκ μέρους των ομάδων. Καταρχήν ο Τόμας Μάνς για τον οποίο θα ισχύσει ο κανόνας του 1,5 λεπτού ομιλίας και μάλιστα πολύ αυστηρά. Ευχαριστώ πολύ. Θα είμαι πολύ σύντομο. Καταρχήν θα ήθελα να ρωτήσω το εξή. Κύριε Επίτροπε, υποθέτω ότι θέλετε να κάνετε το διάλογο με εμά. Συμφωνείτε, ναι. Αλλά για να γίνει ένα διάλογο και για να, πει, και για να, λέει, να ισχυρίζεται κανεί ότι Λισαβόνα δεν λειτουργήσε καλά, αλλά χρειαζόμαστε ένα νέο μοντέλο. Ε, για να γίνει κάτι τέτοιο, χρειαζόμαστε χρόνο για να μπορέσει να εισακουστεί η φωνή του Κοινοβουλίου, καθώ και του κοινωνικού εταίρου, του οποίου θέλετε να συμπεριλάβετε για την διαβούλευση σε ορισμένου τομεί. Χρειαζόμαστε την των πολιτών, στρατηγική 2020. Πώς μπορούμε αλλιώς να προσπαθήσουμε να δημιουργήσουμε ένα κοινωνικό μοντέλο. Ε, ε, χρειαζόμαστε ένα τέτοιο μοντέλο συνεργασίας. Πιστεύετε ότι τα κριτήρια τα οποία έχουν διατυπωθεί η κυρία Τσίμερ επεσήμενε το ζήτημα της φτώχειας. Υπάρχει το ζήτημα του, της ποσόστοσης των όσων διακόπτουν το σχολείο. Ε, συμφωνείτε ότι οι χώρες μέλη ε, θα συνεργαστούν ε, σε όλα αυτά. Θεωρείτε ότι θα συνεργαστούν σε όλα αυτά. Και τρίτη παρατήρηση. Η βιομηχανική πολιτική. Δεν χρειαζόμαστε εδώ ένα μέτρο για την επαναβιομηχανοποίηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν θα ήταν ένα σημαντικό βήμα στο οποίο θα έπρεπε να συμβάλλετε κι εσείς κύριε πίτροπε. Η κυρία Τούρινγκ έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ τον κύριο Επίτροπο που ξανά ήρθε στην Επιτροπή μας. Ευχαριστώ πολύ για τη διαφάνεια αυτή. Και όσον αφορά την στρατηγική του 2020, ελπίζω να εξετάσετε την έκθεση της Επιτροπής μας, διότι Εγώ θα ήθελα η ανάπτυξη μιας κοινωνικής Ευρώπης να τεθεί ε, στην ημερήσια διάταξη και δεν ξέρω αν θα το προλάβουμε αυτό μέχρι τον Ιούνιο. Είναι κάτι που μου λείπει όμως και όπως αναφέρθηκε ανησυχώ ότι οι στόχοι που αφορούν την ένδια και οι στόχοι που αφορούν την εκπαίδευση ε, θα ξεχαστούν τελείως. Όσον αφορά το πρόγραμμα εργασίας, θα ήθελα να επενέσω πολλές από τις πρωτοβουλίες. Ένα πράγμα μου λείπει. Βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή σε μεγάλη κρίση και υπάρχει δυνατότητα αναπροσαρμογής. Γιατί η Κομισιόν δεν παίρνει πρωτοβουλία για μεγάλα εγχειρήματα σχετικά. Τι θα κάνουμε με το, τα 23 εκατομμύρια ε, ανέργους, για παράδειγμα. Θα πρέπει να αρχίσετε να τα σκέφτεστε αυτά τώρα, διότι αλλιώς θα συναντήσουμε σημαντικά προβλήματα. Και αυτό δεν το βλέπω στο πρόγραμμα εργασίας πουθενά. Τέλος, ε, μία τελευταία ερώτηση. Πού βρίσκονται οι συγκεκριμένοι στόχοι που βρίσκονταν στις προηγούμενες κατευθύνσεις γραμμές, αν μπορείτε να απαντήσετε. Ο Επίτροπος, ε, τηλεγραφικά. Ε, η έννοια της οικονομικής ανάπτυξης, κατά τη γνώμη μου, είναι σημαντική, είναι στόχος, όχι επειδή πιστεύουμε ότι το ΑΕΠ είναι τέλειος δείκτης ή ότι χρειαζόμαστε την ανάπτυξη χάρη της ανάπτυξης, αλλά επειδή πιστεύουμε ότι αν έχουμε οικονομική ανάπτυξη, αυτό θα δείξει ότι η Ευρώπη αναπτύσσει την ανταγωνιστικότητά της απέναντι στο υπόλοιπο του κόσμου και μας δίνει καλύτερη ευκαιρία να αυξήσουμε την ευημερία ε, τον πλούτο, ε, τη δημιουργία θέσεων απασχόληση και την κοινωνική ένταξη. Κάποιοι από του οικονομικού δείκτε, όπω το ΑΕΠ μπορεί να μην είναι η καλύτερη επιλογή, μπορεί να είναι η δεύτερη καλύτερη λύση μόνο, ε, αλλά πιστεύουμε ότι είναι καλό τρόπο να ακολουθήσουμε την ατζέντα υπέρ τη απασχόλησης και υπέρ τη ανάπτυξη. Και η Κομισιόν συμφωνεί, το Σώμα των Επιτρόπων συμφωνεί πάνω σε αυτό. Η σχέση ε, απασχόλησης και ανάπτυξης είναι ε, ένα δύσκολο θέμα διότι ήδη βλέπουμε κάποια σημάδια ανάπτυξης όσον αφορά το ΑΕΠ. Δεν βλέπουμε όμως να υπάρχει ανάπτυξη αύξηση των θέσεων απασχόλησης ε, στα κράτη-μέλη. Πιστεύουμε ότι αυτό δεν είναι ασυνέπεια, είναι καθυστέρηση στη φάση και θα πρέπει να εργαστούμε σκληρά με όλα τα μέσα που έχουμε, με όλες τις πολιτικές που έχουμε, να χρησιμοποιήσουμε τα χρηματοδοτικά μέσα που έχουμε, για να γίνει ο κόσμος απασχολήσιμος, για να μειώσουμε την καθυστέρηση αυτή ανάμεσα στην ανάπτυξη ε, του ΑΕΠ και την, ανάπτυξη, την ε, δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης γιατί μιλάω για ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, διότι μιλάω όχι μόνο εδώ αλλά και αλλού για την ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Ε, και το κάνω αυτό επειδή, όχι, όχι επειδή πιστεύω ότι θα έχουμε περισσότερα μετρητά όσον αφορά τα νούμερα στο Ταμείο αυτό, αλλά επειδή πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να βελτιώσουμε τη δουλειά, τη λειτουργία του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και μπορούμε να εργαστούμε γρήγορα για να έχουμε πιο αποτελεσματική χρήση του κοινωνικού ταμείου, καθώς και καλύτερη αξιολόγηση η οποία θα βοηθήσει στη δημιουργία ενός καλού κύκλου, όχι φαύλου κύκλου. Επίσης πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να έχουμε καλύτερη συνεργασία με, άλλους, ε, με άλλες πηγές χρηματοδότησης ε, θα συναντηθώ με τον πρόεδρο της ε, Ευρωπαϊκής Τράπεζας ε, Ανάπτυξης για, και έχω μιλήσει και με άλλους ε, πρόεδρους τραπεζών για να βρούμε τρόπους συνεργασίας και να αυξήσουμε το δυναμικό του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Αυτό είναι πολύ σοβαρή δουλειά. Σχεδιάζουμε μια διάσκεψη τον Ιούνιο για το μέλλον του Κοινωνικού Ταμείου και είμαι βέβαιος ότι και η ευρωβουλευτές ε, θα ενδιαφερθούν γι' αυτό και θα ενημερωθούν ανάλογα. Όπως είπα, το ΑΕΠ δεν είναι απαραίτητα ο πιο τέλειος δείκτης, θα πρέπει να το χρησιμοποιήσουμε όμως. Υπάρχει και μια τεχνική συζήτηση σχετικά με τους δείκτες για την ένδια και τη μείωση της ένδια. Αυτό αποτελεί μέρος της, ε, του διαλόγου που έχουμε αυτή τη στιγμή και ε, στα πλαίσια της Κοινωνικής Επιτροπής και αλλού. Ναι, είναι δύσκολο το θέμα. Ναι, η πρώτη αντίδραση μπορεί να είναι επιφύλαξη από κάποιες πρωτεύουσε. Η πρώτη αντίδραση μπορεί να αντικατοπτρίζει κάποια επιφύλαξη από κάποιες ε, πλευρές, όπως άλλωστε και οι πρώτες αντιδράσεις για την ε, επίλυση της κρίσης ε, λόγω έλλειψης κατανόησης του μεγέθους του προβλήματος ε, και την έλλειψη κατανόησης της κοινωνικής κρίσης. Υπάρχει όμως τεχνικός, γίνεται, πραγματοποιείται τεχνικός διάλογος, εργαζόμαστε με βάση μια σειρά δικτών, όχι μόνο αυτούς που είδατε στην ανακοίνωση της Κομισιόν της 3ης Μαρτίου, τον αυτών που αναφέρεται στο 60% για τη φτώχεια. Υπάρχουν ε, όμως και άλλοι δείκτες που μπορεί να αποτελέσουν μέρος μιας λύσης. Και η ηλική στέρηση αναφέρεται και χρησιμοποιείται συχνά στην κοινωνική πολιτική και επίσης εξετάζεται η δυνατότητα εξέτασης των ε, νοικοκυριών ε, που έχει χτυπήσει η ανεργία και προσπαθούμε να βρούμε ποια θα είναι η καλύτερη απάντηση στα ερωτήματα αυτά. Είμαστε πεπισμένοι ότι όταν υπάρξει πολιτική δέσμευση για μείωση της ένδυας ε, στα πλαίσια του προγράμματος Ευρώπη 2020, η δουλειά που θα απομείνει ε, απλά θα είναι η εξέβρεση του πιο κατάλληλου δίκτυου. Η βιομηχανική πολιτική στην οποία αναφέρθηκε ο κύριος Μαν είναι πρωτοβουλία κλειδί στα πλαίσια του προγράμματος Ευρώπη 2020 και πιστεύω ότι θα οδηγήσει σε νέο διάλογο ε, για το ρόλο της βιομηχανίας και της βιομηχανικοποίησης στην Ευρώπη. Και θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη της τις εμπειρίες της τελευταίας 25 ετίας στους διάφορους τομείς της βιομηχανίας. και πιστεύω ότι ο αρμόδιος επίτροπος ε, θα εξετάσει προσεκτικά το θέμα και θα συμβάλλουμε και εμείς όσον αφορά την πτυχή το, της απασχόλησης. Σίγουρα συμφωνώ ότι δεν έχουμε ακόμα κοινωνική Ευρώπη. Έχουμε 80 εκατομμύρια ε, φτωχούς. Το 10% του εργατικού δυναμικού είναι άνεργο. Και σε κάποια κράτη-μέλη είναι κρίσιμη η κατάσταση όσον αφορά την ανεργία των νέων. Δεν βρισκόμαστε λοιπόν σε θέση να πούμε ότι έχουμε μια κοινωνική Ευρώπη. στόχο όμω είναι να ενισχύσουμε την κοινωνική διάσταση του ευρωπαϊκού προτύπου. Υπάρχει συνένεση σχετικά με αυτό και είμαι βέβαιος ότι το πρόγραμμα Ευρώπη 2020 θα μπορέσει να παρουσιάσει θετικά αποτελέσματα. Γνωρίζω τα μέλη και αισθάνομαι πως ζητούν να περιοριστείτε και εσείς στον χρόνο ομιλία σα. Ε, άρα λοιπόν είναι η τελευταία φορά που μιλήσατε όσο θέλατε. Οι επόμενοι ομιλητέ είναι η κυρία Ράπτη, η κυρία Ράπτη και μετά η κυρία Στανού. Ε, ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Υποθέτω ότι το χρόνο που πήρατε από τον κύριο Επίτροπο τον δίνετε σε μένα. Ε, έχω τέσσερις ερωτήσεις, πολύ συγκεκριμένες σας ευχαριστώ που είστε και πάλι εδώ. Ε, εκτός από φρέσκα νέα, θέλω να πιστεύω ότι θα μας δίνετε και φρέσκες απαντήσεις που θα μας αρέσουν και στο μέλλον. Ε, το ένα θέμα που θέλω να ρωτήσω είναι τι γίνεται με τις απολύσεις, διότι μας ρωτήσατε, για, μας περιγράψατε την διάθεσή σας να δημιουργήσετε θέσεις εργασίας. Αλλά ξέρετε, χάνονται κιόλας θέσεις εργασίας. Το δεύτερο έχει να κάνει με την εκπαίδευση. Μας μιλήσατε για νέα κατάρτιση, για νέες δεξιότητες, μας μιλήσατε για νέους που θα έχουν περισσότερα προσόντα. Πριν φτάσουμε όμως εκεί υπάρχουν οι νέοι που βγαίνουν από το σχολείο και αυτούς τους νέους πρέπει να τους κρατήσουμε μέσα στο σχολείο και να τους κάνουμε να τελειώσουν το σχολείο με επιτυχία. Και υπάρχει και το θέμα της φτώχειας. Το θέμα της φτώχειας είναι ένα θέμα που συζητείται όχι μόνο στην Κομισιόν, όχι μόνο στο Κοινοβούλιο, υπάρχει και το Συμβούλιο. Τι γίνεται με το Συμβούλιο και το θέμα της φτώχειας. Merci beaucoup, Madame puis Madame Madame Κύριε Επίτροπε, η Ευρώπη χρειάζεται μια στατική του μέλλοντος και ε, μιλούμε για τις κατευθυντήριες γραμμές για την πολιτική απασχόλησης, ιδιαίτερα για μια πολιτική για την αγορά εργασίας που να δείχνει προς το μέλλον. Νομίζω ότι ο στόχος της πλήρους απασχόλησης είναι κάτι που δεν θα πρέπει να χάσουμε, χάσουμε από τα μάτια μας ε, και θα πρέπει να διατυπώσουμε κάποιους φιλόδοξους μακροπρόθεσμους ε, στόχους. Και νομίζω ότι θα πρέπει πραγματικά να μην παραιτηθούμε από αυτή τη φιλοδοξία. Είπατε ότι θέλετε να δημιουργήσετε θέσει εργασία πάση θυσία. Ή κάπως έτσι το διατυπώσατε. Για μένα, για το μέλλον της εργασίας είναι σημαντικό το, σημαντική μείωση των επισφαλών, της επισφαλούς εργασίας. Λιγότερο χαμηλή μισθή, ε, ε, λιγότερη επισφαλής εργασίας κλπ για μένα είναι επίσης σημαντικό να μην βλέπουμε μόνο μονόπλευρα το πώς ε, μπορούμε να αυξήσουμε τη λεγόμενη flexicurity, αλλά στον τομέα αυτό θα πρέπει... Ε, υπάρχουν διαφορετικές προποθέσεις πλαίσιο στην Ευρώπη. Ε, την άποψή μου ότι εδώ θα πρέπει να δημιουργήσουμε κάποιες προϋποθέσεις πλαίσιο και στις άλλες χώρες μέλη για να εφαρμοστεί η flexicurity. Ευχαριστούμε πολύ. Κυρία Φιγκερέδο. Σας ευχαριστώ. Πολύ ε, σύντομα γίνεται πολλής λόγος για την ένδυα. Εγώ ήθελα να τονίσω ότι Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, 85 εκατομμύρια άνθρωποι ζουν σε κατάσταση φτώχεια εντό τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ίσω και περισσότεροι, αν λάβουμε υπόψη, ότι τα στοιχεία αυτά έχουν φέρουν την ημερομηνία τη 31η Σεπτεμβρίου, ε, Δεκεμβρίου συγγνώμη, 2008 για να βγούμε από αυτή την κατάσταση δεν αρκεί να λέμε ότι θα καταπολεμήσουμε τη φτώχεια. Είναι απαραίτητο να αλλάξουν οι πολιτικές που οδήγησαν σε αυτή την κατάσταση. Και όταν οι χώρες όπως η δική μου αντιμετωπίζουν την ανάγκη να καλύπτουν τα κριτήρια του Συμφώνου Σταθερότητας και άρα να περιορίσουν ε, κάθετα τις επενδύσεις, ε, τις ε, κοινωνικές παροχές ε, και τη βοήθεια για τη δημιουργία θέσεων απασχόληση, το μόνο αποτέλεσμα μπορεί να είναι περισσότερη αυτόχεια. Πώς θα περάσουμε λοιπόν από τη λόγια στην πράξη, ποιε πολιτικές θα χρησιμοποιήσουμε, πότε θα δώσουμε τις δυνατότητες στην κοινωνική βιωσιμότητα και όχι στην οικονομική βιωσιμότητα. σα ευχαριστώ πολύ. Ο κύριο Πουπάκη. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Το πρόγραμμα εργασιών της Επιτροπής αποτελεί τη βάση για μια νέα αναπτυξιακή πορεία με ενίσχυση ανταγωνιστικότητας και ενδυνάμωση κοινωνικής συνοχής. Σε αυτό το πλαίσιο είναι εντελώς απαραίτητο η διασφάλιση διατηρησιμότητας και ενίσχυση των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης των χωρών, όπου όμως για παράδειγμα έτσι, είναι, θα ήταν εξαιρετικά σημαντικό να υπάρχει για τους αυτοαπασχολούμενους παράδειγμα ειδικό νομικό πλαίσιο που θα διέπει τα εργασιακά θέματα που αντιμετωπίζουν οι, αυτοαπασχολούμενοι, όπως και σαφής διάκριση μεταξύ αυτοαπασχολούμενων και μισθωτών, όταν όλοι γνωρίζουμε ότι με το καθεστώς της συγκαλυμμένης απασχόλησης χάνεται ένα μεγάλο μέρος των εργοδοτικών εισφορών για τα συνταξιδοτικά σημεία και μιλάμε για τα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης. Επειδή δεν φαίνεται να περιλαμβάνεται σε αυτό το πρόγραμμα των εργασιών του 2010 κάτι τέτοιο, το ερώτημά μου είναι αν έχει προγραμματιστεί να γίνει μια τέτοια εξέταση αυτών των ζητημάτων. Ευχαριστώ. Monsieur le Commissaire, en minutes, si vous voulez. Κύριε Πίτροπε, 5-6 λεπτά παρακαλώ έχετε. Σας ευχαριστώ. Δεν μπορούμε να εμποδίσουμε όλες τις πωλήσει. Η Κομισιόν έχει μια στρατηγική να βοηθήσει στην μετάβαση, να βελτιώσει την απασχολησιμότητα και να βελτιώσει την ασφάλεια της απασχόλησης για όσους την έχουν. Τα μέσα που χρησιμοποιούμε, χρησιμοποιούμε μάλλον κάθε δυνατό μέσο για αυτή την κατεύθυνση, προς αυτή την κατεύθυνση. Βέβαια δεν, μπορώ, δεν μπορούμε παρά να ε, διαπιστώσουμε ότι βρισκόμαστε σε προχωρημένο στάδιο όσον αφορά την αναδιάρθρωση. Δυστυχώ οι απολύσει είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε να χειριστούμε, διότι αυτό είναι κομμάτι της των οικονομικών εξελίξεων. Ε, Όπω δημιουργούνται θέσει απασχόληση, έτσι καταργούνται κιόλα. Εμεί θέλουμε να βελτιώσουμε την ισορροπία και να έχουμε περισσότερε θέσει που δημιουργούνται από αυτέ που καταργούνται. Και βέβαια τα τελευταία δύο χρόνια ε, τα πράγματα ήταν αντίθετα. Γνωρίζετε πολύ καλά το τοπίο, δεν χρειάζεται να σας εξηγήσω το γιατί. Τώρα, για τους νέους, είναι σαφές ότι αυτό που εκφράζουμε στην ε, Στρατηγική Ευρώπη 2020 είναι αυτό, το να ενθαρρύνουμε τους νέους ώστε να παραμείνουν ε, στην εκπαίδευση για να μπορέσουν να κερδίσουν ε, πιο χρήσιμη και πιο σοβαρή επαγγελματική κατάρτιση δεν έχει να κάνει μόνο με την αύξηση του ποσοστού των όσων ε, έχουν πανεπιστημιακά πτυχία, αν και αυτός είναι και ένας από τους τίτλους ε, στόχους, αλλά θέλουμε να ενισχύσουμε τη δέσμευσή μας για ενίσχυση της ε, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Πιστεύω λοιπόν πως Έτσι απάντησα στην πρώτη ερώτηση. Επίσης, δεν θυμάμαι αν είπα ακριβώς ε, δουλειές με κάθε κόστος, αλλά θέσεις με κάθε κόστος. Πάντως σίγουρα είπα ότι θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να βελτιώσουμε, να αυξήσουμε τον αριθμό των νέων θέσεων. Υπάρχουν δύο χωριστές κατευθυντήριες γραμμές. Η μία είναι για την ποσότητα και η άλλη είναι η 7 που... Όχι, οι 8 που αφορά την ποιότητα των θέσεων. Μιλάει για οικονομία που βασίζεται στη γνώση, μιλάει για την, την βελτίωση του περιεχομένου της γνώσης, αυτό δεν αναφερόταν χωριστά στην ε, Στατηγική Ευρώπη 2020, αλλά εδώ αντικατοπτρίζονται και οι δύο αυτές ε, πτυχές και, και στις κατευθύντερες γραμμές αναφέρονται χωριστά με, με την ίδια έμφαση. Τώρα δεν μπορούμε να βρούμε χωριστές, ε, μάλλον μαγικές συνταχές για όλα τα κρατημέλη. Αντίθετα μάλιστα όσον αφορά την θέση και την μείωση της φτώχειας τα κράτη-μέλη θα πρέπει να αναπτύξουν τα δικά του προγράμματα ανάλογα με τι ιδιαίτερε του ε, συνθήκε. Γιατί οι προκλήσει μπορεί να είναι πολύ διαφορετικέ στην Ισπανία από ό,τι στην Ολλανδία, από ό,τι στο Ηνωμένο Βασίλειο και τη Ρουμανία, α πούμε. Δεν μπορεί να υπάρξει λοιπόν ομοιόμορφη προσέγγιση. Θα πρέπει να είναι κάθε φορά κομμένη και ραμμένη στα μέτρα του κάθε κράτους με συμμετοχή του ίδιου του κράτους μέλους κάθε φορά. Αλλά από τη στιγμή που βλέπουμε τη δέσμευση του κράτους μέλους για να αποδώσει σε αυτούς τους στόχους θα μπορούμε να το βοηθήσουμε με βάση τα μέσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και επίση, δεν μιλάμε μόνο για οικονομική σταθερότητα και βιωσιμότητα, γι' αυτό και στοχεύουμε στην μείωση τη στόχε και σε όλες τις ομάδες τις ηλικιακέ, εκτός δηλαδή του εργατικού δυναμικού. Μιλάμε και για τους ηλικιωμένου και για τα παιδιά και με τη Βελγική Προεδρία συνεργαζόμαστε για την μείωση της στόχης, ιδιαίτερα για τη μείωση της στόχης των παιδιών. Και αυτό θεωρούμε πως είναι θέμα κλειδί για την κοινωνική βιωσιμότητα και απασχολησιμότητα των επομένων γενεών. Και όσον αφορά τους ηλικιωμένους, στο πράσινο βιβλίο θα ξεκινήσουμε, μια, θα δώσουμε μάλλον λαβή για μια ευρύτερη συζήτηση όπου θα, ε, καλυφθούν πολλά και διάφορα θέματα συμπεριλαμβανομένες της καταλληλότητας των συντάξεων, συμπεριλαμβανομένες της ε, ενεργούς γύρανσης και όλων των πτυχών κοινωνικής ασφάλισης που προκύπτουν και συνδέονται με την κινητικότητα, την δυνατότητα συνταξιοδότησης που θα είναι πολύ δύσκολες συζητήσει, αλλά θα πρέπει δυστυχώς να τις αντιμετωπίσουμε και πολύ σύντομα μάλιστα. Okay. Μάλιστα. Σέρζιο Κομφεράτη και ο κύριος Τούσας μετά στη συνέχεια. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Προεπίτροπε, το 2010 είναι το έτος καταπολέμησης της ένδυας. Η κατάσταση όλο ένα και πιο ανησυχητική είναι. Τα στοιχεία που μας έδινε πριν από λίγο η συνάδελφος Φιγερέδο ήταν για το 2008. Άρα λοιπόν μπορεί κανείς ρεαλιστικά να σκεφτεί πως η κατάσταση είναι ακόμα πιο σοβαρή και δύσκολη. Και σας ρωτώ το εξή. Δεν θεωρείτε ότι το ελάχιστο εισόδημα κατάλληλο για ολόκληρη την Ένωση, προσαρμοσμένο για ολόκληρη την Ένωση θα μπορούσε να αντισταθμίσει τη φτώχεια και κυρίως αν από πλευρά της Κομισιόν υπάρξουν δράσεις προς αυτή την κατεύθυνση. Γιατί με βάση τα όσα εσείς εγκρίνατε, ε, αόριστα και γενικά μου φαίνονται όλα αυτά. Η περάσπιση των εισοδημάτων, εντάξει, είναι μια ανακοίνωση, μια εξαγγελία καλών προθέσεων. Όμως εγώ πιστεύω θα πρέπει να υπάρχουν δεσμευτικά και λειτουργικά μέσα, ε, όπως ας πούμε ένα ελάχιστο εισόδημα για ολόκληρη την Ένωση. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Τούσας. η εκτίμηση που περιλαμβάνεται στην εισαγωγή του προγράμματος της Επιτροπής για το 2010 ότι δήθεν η Ευρωπαϊκή Ένωση συνειδητοποίησε τις σχέσεις αλληλοεξάρτησης που την χαρακτηρίζουν και ένωσε τις δυνάμεις της για να αντιμετωπίσει την κρίση κατά την άποψή μου είναι σε πλήρη αναντιστοιχεία από την πραγματικότητα από τις σύγχρονες ανάγκες της εργατικής λαϊκής οικογένειας. Και αυτό αποδεικνύεται από την ίδια τη ζωή. Αν κάποιος ανατρέξει στο μηχανισμό, το μειχτό μηχανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στην Ουγγαρία, στη Λετωνία, στη Ρουμανία, οι ανακοινώσει σε ό,τι αφορά την Ελλάδα θα δει σκληρά αντιλαϊκά μέτρα που υποθηκεύουν για γενναίες το μέλλον και τη ζωή των εργαζόμενων σε αυτές τις χώρες και όχι μόνο. Αφού τα τύμπανα πλέον χτυπούν και επιδρούν ως ντόμινο και για μια σειρά άλλες χώρες κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό πρέπει να αποτελέσει σαν κόκκινο νικλωστή και να αποτυπωθεί στο μυαλό πολιτικό, ως ένα βασικό πολιτικό συμπέρασμα για όλους μας. Γνωρίζουμε που βρισκόμαστε, έτσι λοιπόν... Συνάδελφε, ευχαριστώ. Κύριε Κόζα. Θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας σε τρεις τομείς. Και θα είμαι σύντομος. Καλωσορίζω αυτό που είπατε, ότι θα υπάρξουν μελέτες επιπτώσεων και αναλύσεις. έτσι ώστε να εξομαλυνθεί η νομοθεσία. Η, κατά το, πολιτική κατά το διακρίσεων έχει καθυστερήσει εδώ και δύο χρόνια. Ίσως θα είναι καλό ε, θέμα για μια ανάλυση των επιπτώσεων. Στι πρωτοβουλίε πάντω Φλέξ, εγώ θέλω να σα προτείνω να λάβετε υπόψη τα άτομα με ειδικέ ανάγκε. Γιατί αν δεν τα λάβετε υπόψη, δεν θα δοθούν λύσει για τα άτομα αυτά. Έπειτα, υπάρχει ένα κενό το οποίο θα πρέπει να καλυφθεί σε σχέση με τα θεμελιώδη δικαιώματα και τον χάρτη. Στο πρόγραμμα εργασίας δεν αναφέρονται καθόλου τα άτομα με ειδικέ ανάγκε. Αναφέρεται την ομάδα των γυναικών, αναφέρεται την ομάδα των Ρώμα, αλλά όχι τα άτομα με ειδικέ ανάγκε και θα πρέπει να αναφέρονται συγκεκριμένα. Σας ευχαριστώ. κυρία Πλούμ. Ευχαριστώ τον Επίτροπο για την έκθεσή του και για τις διευκρινήσει του. Συμφωνώ απόλυτα με το γεγονό ότι το έτο 2010 είναι εξαιρετικά σημαντικό καθώ είναι το έτο κατά πολέμηση στόχες. Είναι όμω επίση, το θέμα, ή μάλλον το έτο όπου προβλέπουμε με τι θα μοιάζει η αγορά εργασίας το 2015 και το 2020. Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας σε μια πτυχή. Η Ρουμανία και η Βουλγαρία είναι οι χώρες που μπήκαν τελευταίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ξέρω πως τα δικά μας πρότυπα και προγράμματα όσον αφορά την αγορά εργασίας είναι διαφορετικά. Αλλά Προσπαθώ να πιστέψω ότι θα στρέψετε το βλέμμα σας και στους ε, περιορισμούς που υπάρχουν στην αγορά εργασίας σε εννέα κράτη-μέλη εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης περιορισμούς που επιβάλλονται στις χώρες ε, ρουμανικής και βουλγαρικής προέλευσης. Και ήθελα να σας ρωτήσω κύριε Επίτροπε, αν στο διάλογό σας με τα κράτη-μέλη στις διάφορες ε, ειδικέ επιτροπές της Κομίσιον κατά τη διάρκεια των συζητήσεών σας με τις κυβερνήσεις των κρατών μελών ε, θα μιλήσετε η πρόεδρος διακόπτη για αυτούς τους περιορισμούς έναντι των Βούλγαρων και Ρουμάνων εργαζομένων που μπήκαν Πρώτου 2007 στην Ένωση. Ευχαριστώ. Uh, Η κρίση αυτή δεν είναι κάτι που βλέπει κανείς κάθε μέρα. Και δεν μπορούμε να αξιολογήσουμε τις εμπειρίες των τελευταίων δύο ετών ως αν ε, πρόκειται για κανονικές διαδικασίες ε, και να μπορούν τα ε, διάφορα, να μπορούν διάφοροι φορείς να εργαστούν κανονικά. Η κρίση αυτή κάθε μήνα μας φέρνει νέες εκπλήξεις και νέες προκλήσεις. Είναι σαφές ότι ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτε τα θεσμικά όργανα, ούτε οι εθνικές κυβερνήσεις ε, ήταν προετοιμασμένα να αντιμετωπίσουν κάτι τέτοιο. Αυτό θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη. Τώρα πια όμως Έχουμε δει το βάθος της κρίσης και την επίδρασή της όσον αφορά την απώλεια θέσεων απασχόλησης. Γι' αυτό επιμένουμε στις πρωτοβουλίες μας και στους ποσοτικούς στόχους του 2020. Συμφωνούμε απόλυτα με τις παρατηρήσεις που έγιναν ότι ό,τι αποφασίσουμε τώρα, ο τρόπος που θα ενορχιστρώσουμε την έξοδο από την κρίση, είναι κάτι που θα αποφασίσει, που θα καθορίσει την οικονομική ανάπτυξη της επόμενης δεκαετία. Υπάρχουν τομεί όπου ήδη έχουμε ισχυρά μέσα. Υπάρχουν τομεί όπου ακόμα σε συνεργασία με τα κράτη-μέλη ετοιμάζουμε το θεσμικό πλαίσιο για το προσεχές χρονικό διάστημα. Θα πρέπει επίσης να καταλάβουμε ότι η επικουρικότητα θα συνεχιστεί σε κάποιους τομείς όπως για παράδειγμα για τους βασικούς μισθούς. Φυσικά μπορούμε να εκφράσουμε θέσεις για το θέμα αυτό. Και όπου έχουμε δει να υπάρχει κάποιος κατώτερος μισθός, είδαμε θετικά αποτελέσματα, αλλά δεν μπορούμε, αν σκεφτούμε ρεαλιστικά, να επιβάλλουμε κάτι στα κράτη-μέλη στον τομέα αυτών. όσον αφορά τα άτομα με αναπηρίες και τη σχέση του με την αγορά εργασίας. Πιστεύω ότι αυτό παίζει ρόλο κλειδί στην ε, κατευθυντήρια γραμμή 7 για την απασχόληση και την ανάπτυξη. Ε, στα πλαίσια του 2020 θα πρέπει να δώσουμε ένα συνολικό νούμερο, το 75%. Έχουμε όμως και μια πιο αναλυτική εικόνα και γίνεται πολιτικός διάλογος για να εγκριθούν οι στόχοι, αλλά ξέρουμε ότι ποτέ δεν θα πετύχουμε το 75% εάν δεν αυξήσουμε την απασχόληση σε κάποιες ομάδες, τις γυναίκες, τους πιο ηλικιωμένους και τα άτομα με ειδικές ανάγκες, με αναπηρίες. Έχουμε λοιπόν παραδείγματα χρήσης του κοινωνικού ταμείου για βελτίωση την, ε, της πρόσβασης ανθρώπων με ε, αναπηρίες θα συνεχίσουμε να το χρησιμοποιούμε. Όσον αφορά την καταπολέμηση των διακρίσεων, μαζί με τη Vivian Redding πρέπει να εργαστώ πάνω στο θέμα αυτό. Συνεργαζόμαστε και στενά με το Ινστιτούτο της Βιέννης, το οποίο έχω επισκεφτεί. Όσον αφορά τις χώρες που προσχώρησαν το 2004, ξέρω ότι ε, οι χώρες αυτές επιβάλλουν κάποιους περιορισμούς, ιδιαίτερα Βουλγαρία-Ρουμανία ιδιαίτερα όσον αφορά τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία. Πιστεύω όμω ότι έχουμε ωφέλη από την κινητικότητα του εργα... εργατικού δυναμικού. Ε, την Παρασκευή θα δείτε στην Frankfurter Allgemeine Zeitung ε, άρθρο όπου αναπτύσσω το θέμα αυτό και όταν του χρόνου σταματήσουν οι μεταβατικές διατάξεις θα μελετήσουμε προσεκτικά τον αντίκτυπο και θα χρησιμοποιήσουμε τα αποτελέσματα για να πείσουμε τα κράτη-μέλη ότι θα πρέπει να αρθούν οι περιορισμοί για τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, διότι ειλικρινά δεν περιμένουμε σοβαρές ε, ανατροπές όταν η Γερμανία και η Ουγγαρία ε, σταματήσουν τις μεταβατικές ε, διατάξεις. Thank you very much. Ευχαριστώ η κυρία Κούνς. Ε, κύριε Πίτροπε, έχω δύο συγκεκριμένες ερωτήσεις. Μάλλον μια υπενθύμηση ή ένα αίτημα. Όταν ε, διαπραγματευτήκαμε το, μικροοικονομικό μέσο, ε, εξετάσαμε την πρόοδο που είναι ένα από τα μέσα στα χέρια σας για την εφαρμογή των στρατηγικών σας. Υπήρχε ανακοίνωση της Επιτροπής ε, ότι θα υποβάλλεται πρόταση για τον προϋπολογισμό 2011 με 2013 που θα επιτρέψει την επιστροφή 30 εκατομμυρίων από το απόθεμα ε, στο, ε, να συμπεριληφθεί στο πρόγραμμα Progress. θα ήθελα παρακαλώ να με διαβεβαίωσετε σχετικά με αυτό. Η άλλη ερώτηση είναι ότι αναφερθήκατε στην αξιολόγηση αντικτύπου επανειλημμένα. Εάν θέλουμε να μειώσουμε την ένδια, σημαντικό θα είναι ότι το Ταμείο Συνεχής μπορεί να επηρεάσει τη θέση των Ρώμα στην κεντρική και ανατολική Ευρώπη, αλλά όχι μόνο εκεί. Θα ήθελα να σας ρωτήσω εάν προβλέπετε συγκεκριμένα ε, μέτρα. Είναι λεπτό το θέμα, αλλά είναι πολύ σημαντικό. Ευχαριστώ η κυρία Μωρά και κατόπιν η κυρία Γιασλοβίσκα. Παρακαλώ. Κύριε Πίτροπε, όλοι εδώ θέλουμε να καταπολεμήσουμε την ένδια, να κινητοποιηθούμε για την ανάπτυξη της απασχόλησης. Εσείς ε, ιδιαίτερα αναφέρατε πως θα πρέπει να έχουμε περισσότερους φοιτητές. Επιτρέψατε μου να σας ρωτήσω πώς και τι έχετε προβλέψει ώστε οι φοιτητέ που έχουμε στα πανεπιστήμια να πετυχαίνουν περισσότερο. Σήμερα έχουμε περίπου 40% νέων που βγαίνουν από τα πανεπιστήμια χωρίς να έχουν πτυχίο στο τέλος της δεύτερης ε, χρονιάς σπουδών. Η επιτυχία λοιπόν των ε, φοιτητών στα πανεπιστήμια είναι κάτι πολύ σημαντικό για την ενσωμάτωσή τους ε, στην επαγγελματική ζωή. Τι προτίθεται να κάνει η Κομισιόν, τι έχει προβλέψει. Σας ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Γεσλοβιέσκα. Επίτροπε, απαριθμίσατε ένα σωρό προγράμματα για το 2010, αλλά και καταλαβαίνω ότι είναι πολύ ευκολότερο να σχεδιάζει κανείς παρά να εφαρμόζει. Γι' αυτό θέλω να ρωτήσω, ποια μέσα. Ποιε δράσεις θα έχουν την προτεραιότητα όσον αφορά κυρίω τη βελτίωση των εκπαιδευτικών συστημάτων των κρατών μελών. Επίση, τι ρόλο θα παίξει η ανοιχτή μέθοδο συντονισμού στο πεδίο τη κοινωνική πολιτική καθώς και τι είδου εθνικά προγράμματα περιμένετε όσον αφορά την κοινωνική ολοκλήρωση. Ευχαριστώ. Κυρία Πρόεδρε, αξιότιμα κύριε Επίτροπε, Αναφερθήκατε στην οδηγία για τον χρόνο εργασίας και είπατε ότι προτίθεται να τον κάνετε αντικείμενο επεξεργασία. Διαπίστωση παριθμών 1. Χαιρετίζω εξαιρετικά το γεγονό ότι θέλετε να συμπεριλάβετε τη διαβούλευση με του κοινωνικού εταίρου στην Ευρώπη. Ερώτηση παριθμών 1. Γιατί όμω απαλή εξαιρέσατε από τη διαβούλευση το πιο σημαντικό θέμα, το ζήτημα του opt-out. Χτες είπατε στον τύπο ότι θέλετε να θέσετε στο επίκεντρο της δραστηριότητά σας τον ε, περιορισμό του ανώτατου χρόνου εργασίας. Θέλετε να μας πείτε περισσότερα πράγματα σχετικά. Τρίτον, όσον αφορά το ερώτημα της κυρίας Στάινρουκ εν σχέση με την ανάγκη μόνιμης απασχόλησης. Δεν απαντήσατε αυτή την ερώτηση. Απαντήστε σε μένα αυτό το ερώτημα την περασμένη εβδομάδα, αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να απαντήσετε ο ίδιος συγκεκριμένα το ερώτημα της κυρίας Στάινρουκ τώρα. Ελπίζω ότι ο Επίτροπος ε, θυμάται ποιο είναι το ερώτημα της κυρίας Στάινρουκ που καλείται τώρα να απαντήσει. <laughs> Ναι, όσον αφορά το μικροοικονομικό μέσο, τη μικροοικονομική διευκόλυνση, ε, τα καλά νέα είναι ότι ο προπολογισμό που εγκρίθηκε σήμερα για την Επιτροπή υπάρχει ένα αρκετό περιθώριο. Συνεπώς λοιπόν έχει ληφθεί αυτό υπόψη στο, μετρήτηλο. Ένα αλφα, 7 εκατομμύρια ευρώ προβλέπονται που θα δώσουν αρκετό περιθώριο στο κοινοβίλιο για να εκπληρώσει αυτή την υπόσχεση εν σχέση με την επιστροφή ε, των ε, ποσών αυτών. Όσον αφορά τη χρηματοδότηση των προγραμμάτων για τους Ρωμά, αυτό συζητήθηκε στην Κόρδοβα, στην κορυφή για τους ε, Ρώμα πριν από μερικές μόνο εβδομάδες. Και ε, το εκτιμήθηκε το Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης παίζουν σημαντικό ρόλο όσον αφορά την υποστήριξη της κοινότητας των Ρώμα και την απασχόληση των Ρώμα και την ενίσχυση της εκπαίδευσής τους. Παρ' όλα αυτά θα ήθελα να σε επισημάνω το γεγονός ότι ε, προγράμματα, δεν είναι να συμμαθούν κάποια προγράμματα ε, βάσει ενός εθνοτικού κριτηρίου. Ε, αυτά είναι δυνατή η υποστήριξη της κοινότητας των Ρώμα γιατί συνιστά μια προτεραιότητα της πολιτικής μας και πιστεύω ότι η συνάντηση αυτή κορυφή, στην οποία συμμετείχε και η κυρία Ρέντινγκ και εγώ ίδιος, εκεί ε, θεωρήσαμε ότι η ανακοίνωση αυτή είναι μια καλή ε, πρωτοβουλία και σε αυτή τη βάση μπορούμε να υποστηρίξουμε περαιτέρω προγράμματα για την καλύτερη ενσωμάτωση συγγνώμη, των Ρώμα ε, κάτι που συμβάλλει και στη μείωση της ένδυας στις χώρες όπου υπάρχουν ισχυρές κοινότητες, πολυάριθμες κοινότητες Ρώμα και είναι πέντε αυτές οι χώρες μέλη. Τώρα ε, υπάρχουν ορισμένες ερωτήσεις όπου εμπίπτουν και σε αρμοδιότητα της κυρίας Βασιλείου. Ε, το ζήτημα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης είναι ξεκάθαρα ένα τομέα όπου και οι δύο ε, ενεχόμεθα. Το ζήτημα της αύξησης συμμετοχή στην υψηλή εκπαίδευση σχετίζεται με τη διαπίστωση ότι στην περίοδο της κρίσης αλλά και γενικότερα άνθρωποι που έχουν υψηλότερο επίπεδο εκπαίδευση έχουν περισσότερες πιθανότητες να κρατήσουν τις θέσεις εργασίας ή να αποκτήσουν νέα, μια νέα θέση εργασίας. Υπάρχει σαφώς μια διαφορά μεταξύ ομάδων, ανθρώπων ε, σε συνάρτηση με το επίπεδο εκπαίδευσής τους εκείνοι που δηλαδή εγκαταλείπουν το σχολείο στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, είχαν πολύ αρνητικές εμπειρίες τα τελευταία δύο χρόνια. Πιστεύω λοιπόν ότι στο επίπεδο των αριθμών ισχύει ότι άνθρωποι που έχουν υψηλό μορφωτικό επίπεδο έχουν περισσότερες πιθανότητες να διατηρήσουν την, την θέση εργασίας τους ή να αποκτήσουν μια άλλη θέση εργασίας εφόσον ε, χάσουν την παλιά. Όσον αφορά το χρόνο εργασίας, αυτό που είπα στον τύπο είναι ότι υπάρχει ένα σκεπτικό για τη διατήρηση της ισχύς της νομοθεσίας όσον αφορά το χρόνο εργασία για λόγους υγιεινή και ασφάλεια. Βρισκόμαστε σε μια πρώιμη φάση της διαβούλευση με του κοινωνικού εταίρου και είναι κάπως πρόημο, συγγνώμη, να προβλέψουμε κάποιες ε, λεπτομέρειες εν σχέση με την έκβαση αυτή της ε, διαβούλευση ή εν σχέση με τις λεπτομέρειες της ε, πρότασης που θα κατατεθεί. Το ζήτημα του opt-out δεν ήταν, ε, νομίζω δεν αποτελούσε ερώτηση. Αλλά δεν έχει εξαιρεθεί από τη συζήτηση με τους κοινωνικούς εταίρους. Ίσως θα θυμάστε ότι το είπα στην ακρόαση. Αλλά όταν προτείνουμε κάποια νομοθεσία, η βασική προσέγγιση δεν είναι να προτείνουμε κάτι από το οποίο θα εξαιρεθούν οι χώρες η μία μετά την άλλη. Επιθυμούμε μία νομοθεσία η οποία να είναι εφαρμόσιμη στις περισσότερες εάν όχι σε όλες τις χώρες μέλη. Όσον αφορά τη βιωσιμότητα της εργασίας, κάτι το οποίο συζητήσαμε στο παρελθόν σχετίζεται με το θέμα της προσωρινής ε, σε σχέση σύγκριση με τη μόνιμη απασχόληση. Και αυτό το οποίο είχα πει τότε είναι ότι για τους νέους θα πρέπει να προσπαθήσουμε να μειώσουμε την αναλογία των προσωρινών συμβάσεων γιατί ε, δεν πρέπει να υπάρχει να, να μεσολαβεί ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα μεταξύ τέλους της εκπαίδευσης και απόκτησης μιας μόνιμης θέσης εργασίας, κάτι που συμβαίνει όμως πολύ συχνά στην Ευρώπη. Και αυτό είναι αποτέλεσμα πολλών ερευνών. Θα πρέπει να μπορέσουμε να πετύχουμε ένα επίπεδο μόνιμης απασχόλησης πιο γρήγορα. Ευχαριστούμε κύριε Επίτροπε. Ε, ε, η κυρία Καρίμα Ντελή. Ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε που παρήσαστε εδώ. Εγώ έχω πολλές ερωτήσεις που θα θέσω τάχη. Είπατε ότι θα πρέπει να δημιουργήσουμε απασχόληση και να μειώσουμε την ανεργία. Εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει καταρχήν να επενδύσουμε στην επαγγελματική κατάρτιση. Εκεί ε, αυτές είναι οι βάσεις της ε, μελλοντικής απασχόλησης. Για παράδειγμα, όσον αφορά την θέρμανση του πλανήτη τα κτίρια είναι 40% υπεύθυνα για τα αέρια των θερμοκηπίων. Για να μπορέσει να υπάρξει μια ανακαίνιση των κτιρίων θα πρέπει να υπάρξει εκπαίδευση νέων αρχιτεκτόνων, μαστόρων κλπ. Αυτά, αυτές είναι οι ευκαιρίες απασχόλησης στις οποίες θα πρέπει να επενδύσουμε. Αυτό είναι το πρώτο. Η δημιουργία θέσεων απασχόλησης σημαίνει, συνεπάγεται ότι χρειαζόμαστε μόνιμη απασχόληση. Ε, εσείς το σχετίσετε με την ε, ανάπτυξη. Όταν λέτε ανάπτυξη στις συνθήκες εργασίας, είναι ανάπτυξη βάσει ανταγωνισμού. Άρα ασκείται πίεση στους εργαζόμενους, στους μισθετούς, άρα έχουμε περισσότερο στρες στην εργασία, επαγγελματικέ ασθένειες κλπ. Άρα τι θα γίνει, θα πρέπει να πιέσουμε τους εργοδότες να είναι πιο ευγενικοί με τους εργαζόμενους. Δεύτερον, το δεύτερο ερώτημα αφορά το έτος της ε, καταπολέμησης της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. Εγώ διάβασα πολλές μελέτες που οδηγούν στην εξή διαπίσωση. Οι πλούσιοι γίνονται όλο και πιο πλούσιοι και οι φτωχοί γίνονται όλο και πιο φτωχοί. Πώς λοιπόν προτίθεστε να ρυθμίσετε αυτή την απόκληση. Θα εμπνευστείτε από την ε, εργασία του κυρίου Στίκλιτς, από τους δείκτες που έχει διατυπώσει. Η κυρία Χάρκιν. Ευχαριστώ Πρόεδρε και καλώς ορίσατε Επίτροπα. Είμαι ευτυχής που βλέπω ότι έχετε μια δέσμευση για τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης με την απασχόληση για τους νέους και την ατζέντα για νέες δεξιότητες και θέσεις. Γιατί κάποιε φορέ επικρατεί εντύπωση πως η Ευρωπαϊκή Ένωση και ορισμένε χώρε είναι τόσο απασχολημένε να διορθώσουν τα χρηματοπιστωτικά τους ε, θεσμικά όργανα που δεν ασχολούνται με τον κόσμο. Εγώ πρωτοέρχομαι από μια χώρα που αυτό κάνει αυτή τη στιγμή από ό,τι φαίνεται, αλλά πραγματικά υπάρχει μια ανάγκη να δείξει η Ένωση πως ασχολείται με το προβλήματα του κόσμου και τις ε, δουλειές για τον κόσμο υπάρχει τώρα χάσμα μεταξύ της ανάπτυξης του ΑΕΠ και της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης και ότι διανύουμε μια μοναδική κρίση αυτή τη στιγμή και πρέπει να προσέξουμε και να παρακολουθήσουμε το κενό αυτό γιατί δεν είμαστε βέβαιοι για το πώς θα βγούμε από αυτή την κρίση. Δύο παρατηρήσεις πολύ σύντομες. Είμαι ευχαριστημένη που βλέπετε ε, και εξετάζετε την εφαρμογή του, της οδηγίας για τους αποσπασμένους εργαζόμενους. Υπάρχουν εκεί πολλές αμφισημίες και επίση το γεγονός ότι θέλετε να εξετάσετε το χρόνο εργασίας αλλά και την δημογραφική πρόκληση. Διακόπτη πρόεδρος. Όχι, Πρώμενη ερώτηση θα είναι για την επόμενη φορά. Η κυρία Σλόμπερ και μετά η κυρία Γίδρυξεν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Θα προσπαθήσω να είμαι πολύ σύντομη. Ξέρω ότι κύριε Επίτροπε εργάζεστε ε, για ένα έγγραφο για τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης, πράσινων θέσεων απασχόλησης. Με ενδιαφέρει να μας πείτε πώς περιγράφετε τη διαδικασία μετασχηματισμού και ποιοι είναι οι σημαντικότεροι στόχοι που διατυπώνετε. Δεύτερον, Έρχομαι από μια ομάδα εργασίας όπου η Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Ανάπτυξης ανέπτυξε τις δικές σας ιδέες και κατάλαβα ότι υπάρχουν πολλές αντιπαραθέσεις εν σχέση με την διαμόρφωση της μιας μελλοντική πολιτικής γιατί ε, θέλετε να υποστηρίξετε κάποιες ε, ε, κατευθυντήριες γραμμές ανάπτυξης της πολιτικής απασχόλησης, αλλά δεν θέλετε να χρησιμοποιήσετε τη νομική βάση της πολιτική ε, πολιτικής συνοχής. Μπορείτε να μας το διευκρινίσετε. Η κυρία Γεντρεύσκαγια. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ξέρω πως το όνομά μου δεν είναι εύκολο, αλλά τα πήγατε πολύ καλά. Θα ήθελα να θέσω μια ερώτηση σε σχέση με το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο για την ε, προσαρμογή στην παγκοσμιοποίηση. Είμαι μέλο της Επιτροπής Προπολογισμού και έχω παρατηρήσει ότι αυτή η διαδικασία παραμένει μυστηριώδης και μπορεί να είναι και ανησυχητική. Ότι δηλαδή οι πιστώσει πληρωμών για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο χρησιμοποιούνται ως ένα ορυχείο για τη μεταφορά ε, κονδυλίων προς το Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση. Στην πράξη έχω δει τουλάχιστον 10 από αυτές τις μεταφορές να γίνονται και ρωτώ για... γιατί χρησιμοποιείται το Κοινωνικό Ταμείο για την πληρωμή του Ταμείου για την Παγκοσμιοποίηση και έπειτα Ποιοι είναι οι λόγοι για την εφαρμογή, για, πώς λειτουργεί αυτό το κοινωνικό ταμείο, γιατί κάπως αυτά τα, αυτές οι πιστώσεις φαίνεται να είναι διαθέσιμες. Η τελευταία σας ερώτηση είναι τεχνική. Σε φύση, όπως γνωρίζετε, το Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση είναι ένα σχετικά πρόσφατο καινούριο μέσο και αυτή ήταν η ρύθμιση που βρέθηκε πριν από ένα-δύο χρόνια, ώστε να μην έχει δικό του προπολογισμό στην ουσία το Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση. Είναι κάτι το οποίο σκεφτόμαστε Μήπω θα πρέπει να έχει δηλαδή δική του γραμμή στον προπολογισμό και να μην χρησιμοποιούμε αυτή τη σχετικά περίπλοκη προσέγγιση. Ωστόσο, Υπάρχει και η άποψη ότι εφόσον λειτουργεί σωστά μπορούμε και να το διατηρήσουμε ως έχει. Παρά την περιπλοκότητά του. παρά δηλαδή τον περίπλοκο τρόπο με τον οποίο βρίσκουμε τα κονδύλια και τη στενή σχέση με το κοινωνικό ταμείο. Τώρα, η μεταφορά τη προτεραιότητα από τη χρηματοδότηση των τραπεζών στη χρηματοδότηση των θέσεων, τη δημιουργία θέσεων, Ο τραπεζικό τομέα έπρεπε να σταθεροποιηθεί και έπρεπε να σταθεροποιηθεί μέσω τη επανακεφαλαιοποίηση. Δυστυχώ αυτό ήταν κάτι το οποίο δεν μπορούσαν να αποφύγουν ούτε κυβερνήσει ούτε κανεί. Γιατί διαφορετικά θα είχαν καταρρεύσει τα πάντα. Πιστεύω πως τώρα έχουμε ξεπεράσει αυτή τη φάση και άρα πρέπει να δώσουμε προτεραιότητα στην δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Και αυτό είναι που πιστεύει και η Κομισιόν, το έχει ανακοινώσει σε διάφορες ανακοινώσεις, ενώ ταυτόχρονα θα πρέπει να σχεδιάσουμε μια περίοδο σταθεροποίησης, οικονομικής σταθεροποίησης. Δηλαδή, δεν ήταν μόνο οι τράπεζες που χρειάστηκε να σταθεροποιηθούν μέσω μεγάλων δημόσιων επενδύσεων, αλλά και το πώς θα προχωρήσουμε στην πολιτική δημιουργία θέσεων απασχόλησης, ενώ ταυτόχρονα θα πρέπει να επικρατήσει λιτότητα και σταθερότητα οικονομική. Σε σχέση με τις νέες θέσεις έχουμε κάνει ανακοινώσεις. αλλά έχουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσουμε θέσεις απασχόλησης στον τομέα της ενέργειας, των ε, κατασκευών, στην αυτοκινητοβιομηχανία. Είναι πολύ σημαντική τομή όπου μπορούν να δημιουργηθούν θέσεις απασχόλησης και αθώς και να πρασινίσουν μέσω των επενδύσεων. Να αναφερθώ στι συζητήσει μου με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Έχουμε συντονισμένη προσέγγιση και αυτό είναι και στον ορίζοντα τη Βελγικής Προεδρία. Είναι κάτι πολύ σημαντικό για μας και εργαζόμαστε επί των λεπτομεριών ε, τους επόμενους μήνες. κυρία Ελέν και κυρία Χάρκιν ανέφεραν το θέμα των ηλικιωμένων και των συντάξεων αναφέρεται στο πράσινο βιβλίο αλλά και σε αυτό που ονομάζουμε το δημογραφικό έλλειμμα. Θα επανέλθουμε λοιπόν με τη δημιουργία των λευκών θέσεων όπως λέμε και με καλύτερες πολιτικές για την ε, κοινωνική πρόνοια. Δεν είμαι βέβαιος πως κάλυψα όλες τις ερωτήσεις σας. Uh, in terms of the cohesion framework. Okay, we speak about a regulatory autonomy of... Μιλάμε για μια αριθμιστική αυτονομία του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και, να, και την αποσαφήνιση του ρόλου του. Εγώ προσωπικά δεν λέω πως το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο θα μπορούσε απόλυτα να αποκοπεί από τα υπόλοιπα μέσα, δημοσιονομικά μέσα και επιτρέπως χάνει με τον οποίο συζητώ τακτικά τα θέματα αυτά, ότι έχουμε ένα γενικότερο πλαίσιο πολιτικών συνοχής, έχουμε ένα ισχυρό σύνολο διορθωτικών ταμείων και εντός αυτών θα πρέπει να δώσουμε σχετική αυτονομία σε ορισμένα οικονομικά μέσα δημοσιονομικά μέσα, διότι εξυπηρετούν συγκεκριμένους σκοπούς. Και γι' αυτό και χρειάζεται συγκεκριμένο είδος κανονισμού. Αλλά η στενή συνεργασία νομίζω πως είναι προς το συμφέρον μας και απαιτείται συντονισμός τις λειτουργίες των ταμείων αυτών. Ενώ με μια πλήρη, ένα πλήρη διαχωρισμό κάτι τέτοιο δεν θα ήταν δυνατό. Κύριε Επίτροπε, σε ευχαριστούμε πολύ. Απαντήσατε 23 ερωτήσεις. Υπάρχει ο κύριος Πόντσας Τερόζα και η κυρία Λίνκεβιτς που ήθελαν να υποβάλουν ερώτηση, αλλά έχουμε ξεπεράσει κατά ένα τέταρτο τον προβλεπόμενο χρόνο μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας εδώ. Ε, ωραία, διαμαρτύρεστε, αλλά... Okay. Okay. Don't lose time. Don't lose time, please. Μην χάνετε χρόνο. Δέχεστε να σας υποβάλει μισό λεπτό ο κύριος Πόντσεστε Τε και μισό λεπτό η, η κυρία Μπλένκεβιτς. Δεν ακούγεται, είναι εκτός μικροφώνου. Πώς άνθρωποι έβαλαν το λόγο που δεν, ε, ε, δεν είχαν καν κανένα νεύμα, ενώ εγώ που σας ε, νεύω εδώ και τόση ώρα δεν μου δίνετε το λόγο. Η ερώτηση μου σχετίζεται με τις κοινωνικές υπηρεσίες κοινή ωφέλεια. Είχαμε μια συζήτηση σχετικά τον Επίτροπο εγώ θα προετοιμάσω μια σχετική έκθεση και θα ήθελα να μου πείτε ποια είναι η δική σας προσέγγιση για αυτό το θέμα. Euh, Ευχαριστούμε πολύ. Αλλά θα πρέπει να συγχωρέσετε την ε, γραμματεία, ούτε η γραμματεία, ούτε εγώ σας είδα. Εάν το είχαμε κάνει θα είστε πρώτος. Ε, θα ήθελα να ρωτήσω τον Επίτροπο πώς θα εξασφαλίσει μια ποιοτική απασχόληση για να μειώσει την ένδια. Ποια είναι η δυνατότητα ε, του 10% του κοινωνικού ταμείου για την απασχόληση νέων ανθρώπων και κατά πόσο η πράσινη βίβλος θα καλύψει την, τον οικονομικό κανονισμό για τα ιδιωτικά κεφάλαια. Very telegraphically, yes, yes, yes, yes. Η απάντηση είναι ναι, ναι, ναι, ναι. Ναι. Η πράσινη βίβλος στόχο έχει καλύτερη νομοθεσία και γι' αυτό ο Επίτροπος Μπαρνιέ ε, έχει συνεργαστεί πάνω στο θέμα αυτό μαζί με τον Επίτροπο Ρεν και μένα. Είναι πολύ σημαντικό το θέμα. Δεν βλέπω το θέμα αυτό του 10% διότι σύμφωνα με τις στατιστικές μας το 30% του κοινωνικού ταμείου χρησιμοποιείται με κάποιο τρόπο ε, για τους νέους. Δεν ε, είναι πάντα προφανέ, αλλά αυτό δείχνουν οι στατιστικέ. Όσον αφορά την απασχόληση ποιότητα, έχουμε μία συγκεκριμένη κατευθυντήρια γραμμή και είμαι βέβαιο ότι θα έχουμε πολλέ ευκαιρίε να το συζητήσουμε αυτό. Όσον αφορά τι ε, κοινωνικέ επιχειρήσει κοινή ωφελία, ε, καταλαβαίνω το θέμα αυτό και εκτιμώ ε, αυτό που είπε ο κύριος Στερόσα. Το θέμα είναι ότι βρισκόμαστε σε αρχική φάση του συλλογισμού πάνω στο θέμα αυτό. Θα πραγματοποιηθεί διάσκεψη στη Βαρκελόνη, η οποία και αυτή σχετίζεται με το θέμα αυτό. Και μετά από τη διάσκεψη αυτή τον Ιούνιο θα ακολουθήσει μια περίοδος συλλογισμού διότι είμαι βέβαιος ότι συμμεριζόμαστε τις αρχές, την παροχή ποιότητας, ε, την διασφάλιση της ε, προσβασιμότητας στις ε, δημόσιες υπηρεσίες, στις κοινές υπηρεσίες. Κάτι που ανέφερα και σε προηγούμενη απάντησή μου ε, είναι ότι η ε, περίοδος οικονομικής σταθεροποίησης που θα ακολουθήσει είναι πολύ σημαντική για τις κοινωνικές υπηρεσίες ε, κοινή ωφελίας. Θα πρέπει λοιπόν να επικεντρωθούμε ακριβώς σε αυτή την πρόκληση για να μπορέσουμε να προοδεύσουμε μαζί. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την ευκαιρία πραγματοποίησης της συζήτησης αυτή σήμερα να σας ευχηθώ και καλή συνέχεια. Σας ευχαριστούμε που συνεργαστήκατε μαζί μας. Ε, ελπίζω να πετύχετε καλή νομοθεσία και να ε, έρθετε μόλις έχετε κάτι νέο να μας ανακοινώσετε. Ευχαριστώ πολύ. Αγαπητοί συνάδελφοι, σας προτείνω να περάσουμε αμέσως στο σημείο 7 της ημερήσιας διάταξης. Ε, σας προτείνω να τα εξετάσουμε μαζί το 7 και το 8 γιατί πρόκειται για την προφορική ερώτηση και το σχέδιο ψηφίσματος το οποίο είχαμε προγραμματίσει σε σχέση ακριβώς με τη στρατηγική του 2020 για την οποία θα πρέπει να αποφανθούμε αύριο δεδομένου ότι αυτό το σημείο θα τεθεί στην Ολομέλεια στη Σύνοδο του Μαΐου προς έγκριση μαζί με άλλα κείμενα τα οποία θα εγκριθούν από τις άλλες επιτροπές που έλαβαν σχετικές πρωτοβουλίες. Όσον αφορά την προφορική ερώτηση, η κυρία Λίνη, η αντιπρόεδρός μας, κατέθεσε δύο τροπολογίες που έχουν σαν στόχο να ενισχύσουν τη δέσμευση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη διακυβέρνηση και στη διατύπωση των στόχων ε, θεωρώ ότι είναι τροπολογίες που θα πρέπει να υποστηρίξουμε. Όσον αφορά το ίδιο το ψήφισμα, έχουν κατατεθεί 56 τροπολογίες που ενισχύουν ουσιοδός ορισμένες πτυχές του ψηφίσματος, ιδιαίτερα όσον αφορά τους νέους, τα, ε, τις αναπηρίες ή τις μεθόδους εργασίας που έχουν ε, χρησιμοποιηθεί μέχρι στιγμή ανοιχτές μέθοδοι συντονισμού, καθώς και δύο τροπολογίες τη κυρία Μπιζωτό για τι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και για τη σημασία τη μαθητείας. Όσον αφορά την ουσία αυτών των τροπολογιών, ε, δεν έχω ιδιαίτερα προβλήματα και υπάρχουν κάποιες συμβαστικές τροπολογίες ε, που πρότεινα και νομίζω ότι έχουν εγκριθεί. Αλλά υπάρχει μια τροπολογία του κυρίου Καπρνός, εάν προφέρω σωστά το όνομά του λέει ομιλήτρια, που θεωρώ ότι θέτουν περισσότερες δυσκολίες εφόσον, αφορ... εφόσον προτείνει να επαναθέσουμε το ζήτημα του δημόσιου χρέους ή των δημόσιων οικονομικών σε σχέση ακριβώ με την απασχόληση που έχουν ή να αντικαταστήσουμε στο στόχο της πλήρους απασχόλησης ε, με τον ε, στόχο της λεγόμενης υψηλής απασχόλησης. Είδω λοιπόν τα θέματα. Εγώ είμαι ανοιχτή στη συζήτηση με το σύνολο των συναδέλφων. Κύριε Ορή, έχετε το λόγο. Παρακαλώ. Θα ήθελα να επαναλάβω αυτό το οποίο είπα προηγουμένως, δηλαδή το ΕΛΚ δεν έχει τίποτα κατά αυτό του αιτήματο, αλλά θέλουμε μια γραπτή δήλωση. Και αν υπάρξει μια γραπτή δήλωση, εμείς θα είμαστε κατά. Για να διευκρινίσουμε την κατάσταση, θα ήθελα να προσθέσω ότι όλη η διαδικασία σε σχέση με τη στρατηγική 2020 είναι ταπεινωτική όσον αφορά το Κοινοβούλιο γιατί τα δικαιώματα του Κοινοβουλίου δεν γίνονται σεβαστά, βρισκόμαστε υποπίεση και τρέχουμε σαν τρελή και δεν είναι αξιοπρεπές για το Κοινοβούλιο να αναγκάζεται να αποδεχθεί όλες αυτές τις αποφάσεις και το αποτέλεσμα θα είναι ότι το Κοινοβούλιο υποπίεση ε, θα πει οτιδήποτε και θα δεχθεί σε χαοτικά αποτελέσματα. Εμείς ε, και, και, και όπως σας είπα θα επιθυμούσα να υπάρξει μια γραπτή δήλωση. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Εγώ θα ήθελα με κάθε σεβασμό προς τον κύριο Αρή, Ορή ότι ίσως ε, θα έπρεπε να έχουμε, κάνουμε έναν επιπρόσθετο προβληματισμό. Γιατί συμφωνώ με τα όσα λέει ο κύριος Ορή και έχει κάθε δίκιο να μιλάει για τον ε, ρόλο που καλύτερα να το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που θα ορίσει τα επόμενα δέκα χρόνια το μέλλον της Ευρώπης. Και βρισκόμαστε πραγματικά υποποίηση ενός ε, πολύ βιαστικού χρονοδιαγράμματος και υπάρχουν και οι αποφάσεις των πολιτικών ομάδων που ασχολούνται με ζητήματα απασχόλησης. Όσον αφορά την προφορική ερώτηση, και το ζήτημα του ψηφίσματος. Έχουμε τη δυνατότητα να θέσουμε στο επίκεντρο της ε, συζήτησης το θέμα της απασχόλησης στο πλαίσιο της Ατζέντα 2020 ούτως ώστε να μπορέσουμε με ένα πλατή και γενικό τρόπο να μπορέσει να εισακουστεί η φωνή του Κοινοβουλίου για να δείξουμε στους Ευρωπαίους πολίτες ότι όχι μόνο στις οικογένειες της Ευρώπης το πρώτιστο πρόβλημα είναι η απασχόληση, αλλά και το, η δική μας απόλυτη προτεραιότητα είναι απασχόληση. Θα πρέπει να το κάνουμε σαφές. Γιατί μόνο με τον τρόπο αυτό θα μπορέσει να εισακουστεί και η δική μας φωνή, η φωνή της Επιτροπής Απασχόλησης. Ε, αυτό δεν είναι ένα θέμα το οποίο αφορά τη μία ή την άλλη πολιτική ομάδα, αλλά αφορά το σύνολο του σώματος. Η κυρία Χάρκιν. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Έχω πολύ λίγα να προσθέσω σε αυτά που υπόθηκαν. Γενικά υποστήριζω το θέμα αυτό. Έχουμε κάποια προβλήματα με μία ή δύο τροπολογίες. Υπάρχουν αρκετές ε, τροπολογίες του Μιλάν Κάρμπονα που δεν μπορούμε να ε, στηρίξουμε. Μπορώ να συμφωνήσω όμως με την τροπολογία 15 που λέει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται κυρίως ε, εργατικό, δυναμικό, με υψηλά προσόντα. Ζητήσαμε προφορική τροπολογία στην τροπολογία 9, εκεί που μιλάμε για βασικό στόχο του, της Ευρώπης 2020 θέλουμε να μιλάμε για έναν σημαντικό στόχο αντί για τον κύριο στόχο του, του, της Ευρώπης 2020 και ε, ζητήσαμε και χωριστή ψηφοφορία για την τροπολογία 33 που καλεί την Κομισιόν και το ε, την Κομισιόν και το Συμβούλιο να παρέχουν ε, εγγύηση ε, επαγγελματική, αλλά έχουμε πρόβλημα με ε, το μετά από τέσσερι μήνε ανεργία, διότι αυτό βρίσκουμε ότι είναι υπερβολικά συγκεκριμένο και μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα για τα κράτη-μέλη. Στηρίζουμε δηλαδή το πρώτο μέρο, όχι όμω το δεύτερο. Ε, κατά τα άλλα, ε, με μία ή δύο εξαιρέσει, συμφωνούμε με όλε τι τροπολογίε. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Υπάρχουν άλλοι που θέλουν να πάρουν το λόγο. Εκ μέρους των Πρασίνων να σας ευχαριστήσω για μια πολύ καλή έκθεση. Θα ήθελα να συμφωνήσω με τον κύριο Σέρκας να προβάλλουμε τις θέσεις της Επιτροπής μας. Συμφωνώ και με αυτό που είπε ο κύριος Όρη, ότι ε, πράγματι μπερδευτήκαμε λίγο. Θέλουμε όμως να προωθήσουμε τις ε, θέσεις της Επιτροπής μας. Στηρίζω το θέμα. Ε, πράσινοι υπέβαλαν 20 τροπολογίες, όχι επειδή δεν μα αρέσει το ψήφισμα, αλλά επειδή έχουμε τόσα να προσθέσουμε. Δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες, ε, πολύ σύντομα. Όσον αφορά την εγγύηση για την νεολαία, την τετράμινη, αυτό συμπεριλαμβάνεται αυτή τη στιγμή στι κατευθυντικέ γραμμέ. Ε, τα κράτη-μέλη ήδη δηλαδή έχουν συμφωνήσει πάνω στο ε, τετράμινο. αποτελεί δηλαδή απλά συνέχεια αυτών. θα πρέπει να σκεφτούμε την προφορική τροπολογία, να αλλάξουμε τον κύριο στόχο σε σημαντικό στόχο. Θα το δούμε όμως αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Πόντσια Στερόσα. Σας δίνω πολύ πολύ ευχαριστώ στο λόγο. Ευχαριστώ πολύ και μπορώ να πω τώρα αυτό που ήθελα να πω νωρίτερα. Ευχαριστώ. αυτό που με οδήγησε στο να έχω ανησυχίες όσον αφορά τις ε, προτάσεις της Επιτροπής για το 2020 είναι ότι υπάρχει μια δήλωση στην προσέγγιση τους ότι θεωρούν την πλατφόρμα αντιμετώπισης της ένδυας ως τρόπο διασφάλισης ότι όσοι υποφέρουν αυτό θα μπορέσουν να υποφεληθούν από την ανάπτυξη και τη ε, την δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Δεν υπάρχει όμως καμία ε, ένδειξη εδώ ότι η Επιτροπή θεωρεί την κοινωνική πολιτική συμβολή στην ανάπτυξη ότι η ανάγκη για ισχυρή κοινωνική υποστήριξη αποτελεί προϋπόθεση για την ανάπτυξη των οικονομιών και ότι θα πρέπει οι οικονομίες να αναπτυχθούν με δίκαιο τρόπο και ήθελα να ρωτήσω τον Επίτροπο πώς μπορούμε να διασφαλίσουμε ε, την υπεράσπιση των κοινωνικών υπηρεσιών. Βέβαια, θα ήταν αμέλεια δική μας ε, να μην αλλάξουμε τίποτα στο κείμενο της Επιτροπής. Αλλά πιστεύω ότι αυτό το βασικό θέμα, η βασική παρερμηνία από πλευράς της Επιτροπής την έξοδο από την παρούσα κρίση, αυτό θα πρέπει να συζητηθεί ενδελεχώς ενδεχόμενα σε κάποια άλλη περίσταση. Ο Επίτροπος μίλησε για την κρίση. Το πρόβλημα είναι ότι εκατομμύρια Ευρωπαίων αντιμετωπίζουν την ένδια εφόρου ζωής από τη μέρα που γεννιούνται μέχρι τη μέρα που πεθαίνουν. Και παρόλα τα προγράμματα που είχαμε, παρόλα τα μέτρα, φαίνεται να μην έχουμε μάθει τίποτα σχετικά με το πώ θα αντιμετωπίσουμε το θέμα αυτό. Ευχαριστώ. Ε, για αυτό το σημείο, αγαπητοί συνάδελφοι, θέλετε να έχετε μια ιδιαίτερη προφορική τροπολογία που θα μπορούσε να προταθεί αύριο στην Επιτροπή. Ευχαριστώ πολύ για όλες αυτές τις εισφορές. Στην κυρία Τουρινάν, ε, θα της έλεγα αυτό το οποίο είπα προηγουμένως όταν παρουσίασα την τροπολογία μου. Θεωρώ ότι είναι μια βελτίωση του περιεχομένου του ψηφίσματος και υποστηρίζω τις τροπολογίες. Ε, θα ήθελα να απαντήσω στον κύριο Ορή λέγοντας ότι συμμερίζομαι τις ανησυχίες του που συνδέονται στη μοίρα τη δική σας έκθεσης που από νομοθετική άποψη και από την άποψη αρμοδιότητας αυτής της Επιτροπής είναι πραγματικά η θεμελιωδή, η ουσιαστική έκθεση. Ε, το θέμα όπως εγώ. Εμείς πήραμε μια πρωτοβουλία που επιτρέπει σε αυτό το κοινοβούλιο να είναι σε θέση να εγκρίνει κάτω από ευνοϊκές προϋποθέσεις ή από, ε, ως μη χείρον ε, τις λεγόμενες κατευθυντήριες γραμμές της απασχόλησης. Και αυτή είναι η συζήτηση που είχαμε τους συντονιστές ε, δύο φορές. Ο μηχανισμός ε, ο οποίος λειτουργεί φέτος στους κόλπους αυτού του κοινοβουλίου ε, και βρισκόμαστε σε, μια, σε ένα χρόνο στρατηγικής σημασία όσον αφορά την έγκριση της λεγόμενης στρατηγικής η λειτουργία αυτή είχε κάτι το χαοτικό, απογοητευτικό, γιατί είχαμε την εντύπωση ότι οι προϋποθέσεις εκπόνησης της θέσης του Κοινοβουλίου γινόντουσαν σε γραμμή ζιγ-ζαγ. Δηλαδή ανακαλύπταμε ότι θα έπρεπε να υιοθετήσουμε αυτό το χρόνο το άλλο ή την τάδε μέθοδο της εργασίας ή την άλλη ακριβώς κινούμενη σε ζιγ-ζαγ. Ε, γιατί είχαμε το σχηματισμό της Νέας Επιτροπής, ε, στη συνέχεια ε, τέθηκαν κάποια άλλοι στόχοι και πραγματικά βρεθήκαμε άσχημα προετοιμασμένοι ούτε ώστε να διατυπώσουμε τη θέση του Κοινοβουλίου στην αδικη 2020 κάτω από ευνοϊκές για μας προϋποθέσεις. Οι συντονιστές είπαν ότι θα ήταν ευκταίο ως Επιτροπή Απασχόλησης να μπορέσουμε να αναπτύξουμε τη δική μας άποψη ε, με το πιο οριζόντιο δυνατό τρόπο εν σχέση με την δική μας θεώρηση αυτής της πρώτης στρατηγικής, του 20, της στρατηγικής 2020 από την Επιτροπή. Πιστεύω ότι τέλος ε, υπάρχει μια στιγμή όταν δημιουργείται μια πραγματικότητα θα πρέπει να προσπαθήσουμε εμείς να δούμε τι είναι το πιο αποτελεσματικό έστω και αν δεν ήταν η αρχική μας πρόταση. Και βεβαίω στην αρχή μπορεί κανείς να έχει διαφορετικές ε, θέσεις. Αλλά εμείς ε, κερδίσαμε ε, να έχουμε μια προφορική ερώτηση στην Επιτροπή Απασχόλησης και στη συνέχεια ένα ψήφισμα. Ίσως αυτό δεν είναι το ιδεώδες. Παρόλα αυτά μας επιτρέπει εν σχέση με σημεία που είναι ιδιαίτερα σημαντικά και για τη δική σας έκθεση ήδη από την Άνοιξη να περάσουμε κάποια μηνύματα για θέματα που συζητήσαμε τον κύριο Επίτροπο και που από πολιτική άποψη νομίζω ότι ε, έχουν τη συνένεσή μας, για παράδειγμα, στον αφορά την καταπολέμηση της φτώχειας ή την απασχόληση ή την κατάσταση των νέων. Και θεωρώ κρίμα μια ομάδα τόσο σημαντική όσο το ΕΛΚΕ να μην ε, προσχωρεί σε αυτή την ε, τόσο σημαντική συζήτηση. Ε, ελπίζω ότι ίσως αύριο θα συμφωνήσετε και εσείς μαζί, μα, μαζί μας για να μπορέσουμε να περάσουμε ένα πολιτικό μήνυμα πέρα από αυτές τις ομυρικές μάχες μεταξύ των πολιτικών ομάδων. Έχετε το λόγο. Ναι. Αυτή η πρακτική θα συνεχίσει να ισχύει. Δεν είναι μια έκτακτη κατάσταση. Μετά τη θέση ισχύ της ισχύς της Λισαβόνας, ο καθένας προσπαθεί να πληρώσει το χώρο που του δόθηκε και να εκμεταλλευτεί τη, την ισχύ του. Το Συμβούλιο, η Επιτροπή και το ΕΛΚ. Και νομίζω ότι αυτή θα συνεχίσει να είναι η πρακτική στο μέλλον. Γι' αυτό ε, διαφωνώ με την ε, πρακτική αυτή εσπευσμένων αποφάσεων. Αντί να έχουμε μια σωστή επικοινωνία με το Συμβούλιο και την Επιτροπή. Δεν έχω πρόβλημα με το ίδιο το κείμενο. Το ίδιο το κείμενο είναι σωστό. Αλλά πραγματικά με ενοχλεί αυτό ο τόπος η τεράστια πίεση. Ε, καταλαβαίνω τη θέση σας και νομίζω ότι η διαδικασία που ξεκινήσαμε στο επίπεδο της διάσκεψης των Πρόεδρων της Επιτροπής μας επιτρέπει ακριβώς να εξασφαλίσουμε ότι τουλάχιστον όσον αφορά το συγκεκριμένο ε, θέμα ε, εφαρμογής αυτής της στρατηγικής να βρεθούμε σε μια πιο ευνοϊκή θέση. Σας προτείνω να κλείσουμε αυτό το θέμα της ημερήσια διάταξης το οποίο θα ψηφιστεί αύριο και ενδεχομένως να δούμε γρήγορα τη γνωμοδότηση που θα πρέπει να δώσουμε στην Επιτροπή ΙΝΤΑ εν σχέση με την κοινωνική ευθύνη των εταιριών στις συμφωνίες διεθνούς εμπορίου παρόλο που θα έπρεπε να ψηφίσουμε αυτή τη γνωματοδότηση αύριο και τελικά η ψηφοφορία αναβλήθηκε γιατί ο εισηγητής επί της ουσίας δεν έχει κάνει καταθέσει το κείμενό του. Δηλαδή είναι παράδοξο να εγκριθεί μια γνωμοδότηση για ένα κείμενο το οποίο δεν είναι ακόμα διαθέσιμο. Και αυτό ε, σημαίνει ότι έχει ξεκινήσει ήδη μια συζήτηση και υπάρχει ο εισηγητής Εγώ ευχαρίστω να παρουσιάσω τις τροπολογίες που έχουν κατατεθεί. Επί της ουσία είναι πολύ επικοδομητικές και πηγαίνουν στην κατεύθυνση της πρότασης ψηφίσματος. Εγώ ίδια πρότεινα στους συντάκτες των διαφόρων τροπολογιών ορισμένες συμβαστικές λύσεις τροποποίησης και θα έχουμε την ευκαιρία να ζητήσουμε σχετικά κατά τη διάρκεια της ανταλλαγής απόψεων την 4η Μαΐου. Υπάρχει ένα σημείο το οποίο γύρει πολιτικές αντιπαραθέσεις και είναι επίμαχο. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή υπάρχουν ε, καλές πρακτικές που έχουν αντιπιθεί στον τομέα της κοινωνικής ευθύνης των επιχειρήσεων. Κάποια στιγμή αυτές οι προδιαθέσεις, αυτοί οι κανόνες μπορούν ε, να θεσπιστούν νομοθετικά ούτως ώστε να υπάρξει ένα ίσο επίπεδο εφαρμογής και να, ενισχύσουμε, και να το βάρος αυτών των κανόνων ή προδιαγραφών. Εγώ ε, συζητώ με ορισμένε επιχειρήσεις που εφαρμόζουν αυτό το μοντέλο κοινωνικής ευθύνης. Και φαντάζομαι ότι θα, υπάρχουν, θα βρούμε κάποιες άλλες επιχειρήσεις που αντιτίθενται και έχω την εντύπωση ότι βρισκόμαστε σε μία φάση ανάπτυξης αυτού του μοντέλου όπου θα μπορούσαμε πραγματικά να κάνουμε αυτό το βήμα προς τα μπρος. Ιδού λοιπόν η ουσία των όσων είχα να πω για αυτές τις 50 τροπολογίες που κατέθηκαν για το κείμενο αυτό. Κυρία Βέρχιστρομ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Είναι ενδιαφέρον ότι δεν είπατε να μην έχουμε συζήτηση, αλλά τελικά πρόκειται για συζήτηση, διότι η πρόεδρο παρουσίασε κάποιε γενικέ σκέψεις. Φυσικά είναι σημαντικό ε, η ανάληψη κοινωνική ευθύνη ε, να πραγματοποιηθεί στην ε, κοινωνία. Οι διεθνεί εμπορικέ συμφωνίες είναι παγκόσμιες και επηρεάζουν πολλού. αλλά θα πρέπει οι επιχειρήσει να δουν τους εαυτού του ω κοινωνικού παράγοντε. Σημαντικό όμως είναι να μην νομοθετήσουμε όσον αφορά την κοινωνική ευθύνη. Πιστεύω ότι είναι καλύτερο ε, αν προωθείτε από ανθρώπους που ε, ε, ενδιαφέρονται στις επιχειρήσεις. Δεν πιστεύω ότι πρέπει να επιβάλλουμε περισσότερη νομοθεσία στις επιχειρήσεις. Όπως και η Πρόεδρος έχω συναντηθεί με πολλές επιχειρήσεις στην Ευρώπη που θεωρούν ότι αυτό είναι μεγάλη απειλή και που θεωρούν ότι αυτή την εποχή και υπό το φως ε, της κρίσης ε, να ε, ενσωματώσουμε την κοινωνική ευθύνη στην εμπορική πολιτική χωρίς όμως να νομοθετήσουμε διότι οι επιχειρήσεις ούτως ή άλλως δυσκολεύονται να επιβιώσουν. Τέλος, οι άνθρωποι και οι επιχειρήσεις όπου εργάζονται αποτελούν την τον κοινωνικό ιστό μιας κοινωνίας και αυτά βασίζονται σε θετική οπτική του ανθρώπου και σε θετική οπτική της κοινωνίας και των παραγόντων της. Ε, εδώ λοιπόν υπάρχει η διαχωριστική γραμμή ανάμεσα στην πρόταση αυτή και την ιδεολογία ε, τη δική μου και που έχει παρουσιάσει η Πρόεδρος στο σχέδιο που συζητάμε σήμερα. Ευχαριστώ. Ε, θέλουν άλλοι να πάρουν το λόγο. Ο κύριος Δερόζα. Σε σχέση με το ζήτημα της εταιρική ευθύνη, θα ήθελα να πιστήσω την προσοχή της Επιτροπής στο γεγονός ότι αυτή η Επιτροπή συμμετείχε σε μία ακρόαση σήμερα με την Επιτροπή Ανάπτυξη και την Επιτροπή Εμπορίου για το θέμα της παιδικής εργασίας. Ε, και βεβαίως ε, το θέμα της κοινωνικής ευθύνης τέθηκε στο πλαίσιο αυτό ένα εντυπωσιακό σημείο που ανέκυψε είναι η πολλαπλότητα κριτηρίων που, υπάρχουν σε σχέση με την παρακολούθηση και παλήθευση όσον αφορά τη συμβατότητα με τα κριτήρια του ILO. Ε, και σχέση με τους μη κυβερνητικούς οργανισμούς. ελέγχθη ε, ε, λοιπόν θα πρέπει να υπάρξει μια τυποποίηση αυτών των κριτηρίων και εκτός αν είμαστε και θα πρέπει να ε, είμαστε θα πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη το ζήτημα της εταιρική κοινωνικής ευθύνης από τις εταιρείε. Ορισμένες εταιρείε θεωρούν το θέμα της εταιρική κοινωνικής ευθύνης σαν ένα εργαλείο marketing και το χρησιμοποιούν έτσι ε, και δεν το αντιμετωπίζουν σαν ένα τεράστιο ηθικό ζήτημα. Εάν ε, κάποιοι είναι υπεύθυνοι στο πλαίσιο της, των επιχειρήσεων, θα πρέπει να συνεργάζονται με τη διοίκηση θα πρέπει οι άνθρωποι αυτοί να έχουν αρκετή δύναμη εντός της επιχείρησης ούτως ώστε να προβάλλουν τα θέματα αυτά επαρκώς και να γίνονται και ε, να τους ακούνε. Ευχαριστούμε πολύ. Υπάρχουν άλλες ε, παρεμβάσεις. Όχι, θα ήθελα να σε ευχαριστήσω για την εισφορά σας και το πνεύμα που έγιναν οι παρεμβάσεις σας. Ελπίζω να μπορέσουμε να βρούμε μια συμφωνία στις συνεδρίες της 4ης Μαΐου. Αλλιώς, επί του σημείου αυτού που είναι ιδιαίτερος ε, σημαντικό, όσον αφορά την εκπόνηση μοντέλων κοινωνικής ευθύνης ε, των εταιριών, θα το ψηφίσουμε. Τη Δευτέρα Ιουνίου, βάσει του χρονοδιαγράμματος της Επιτροπής. Ελπίζω ότι μέχρι τότε θα έχουμε το σχέδιο της έκθεσης της Επιτροπή που είναι επί Παραμένουμε σε ένα παρόμοιο σχετικά θέμα, γιατί θα συζητήσουμε τις τροπολογίες, τις συμβιβαστικέ στην έκθεση του συναδέλφου Richard Howitt, που είναι μια γνωμοδότηση της Κομισιόν Ίντα, για την Κομισιόν, για την Επιτροπή Ίντα, για τι κοινωνικέ και περιβαλλοντικές προδιαγραφές στις διεθνείς εμπορικέ συμφωνίες. Είναι μια έκθεση πρωτοβουλία τη επιτροπή ΕΝΤΑ. Κύριε Σιγητά, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Είχαμε τις τροπολογίες κατά την τελευταία ανταλλαγή απόψεων. Δεν χρειάζεται να επαναλάβουμε τη συζήτηση που είχαμε τότε. Ε, απλά θα ήθελα ευχαρίστω να απαντήσω σε οτιδήποτε ε, έχει να ρωτήσει κανείς. Όσον αφορά τους συμβιβασμούς, έχουμε υποβάλει τέσσερις διαφορετικούς ε, συμβιβασμούς στον ε, συνάδελφο Χίκινς ε, που δεν, δεν είμαι σίγουρος αν είναι εδώ. Έχουμε ε, καταβάλει σημαντικές προσπάθειες για να καταλήξουμε σε συμβιβασμό. Δεν θέλω να τον επικρίνω με κανέναν τρόπο, αλλά δεν ήταν δυνατόν με κανέναν τρόπο να καταλήξουμε σε συμβιβασμό με τον οποίο θα ήμασταν και οι ικανοποιημένοι. Ε, ως συντάκτης της προσπάθησα να καταλήξω σε Συμβαστικέ τροπολογίε που πιστεύω ότι θα βρουν την υποστήριξη τη πλειοψηφία τη επιτροπή μα και των περισσότερων ομάδων. Ε, σέβομαι και εκτιμώ τον κύριο Χίγκινς, ε, αλλά δεν μπορώ να στηρίξω τι ε, τροπολογίε του ε, συνολικά. Βέβαια, έχει κάθε δικαίωμα να τι υποβάλει. Όσον αφορά την συμβαστική τροπολογία 1, αυτή έχει να κάνει με την παράγραφο 1, τον ορισμό του δίκαιου εμπορίου, του δίκαι ο κ. Πιτεκιάν ήθελε να συμπεριληφθεί και η αγορά εργασία μαζί με τα δικαιώματα, μαζί με τα συνδικαλιστικά, ε, συγγνώμη, τα εργατικά μαζί με τα συνδικαλιστικά δικαιώματα. Στην παράγραφο 5, όπου αναφερόμαστε ε, με τις ε, μελέτε βιωσιμότητα και αντικτύπου, έλαβα πολύ βοήθεια παρόλο που Ιδανικά δεν θα συμπεριλάμβανα την Λατινική Αμερική. Θα στηρίξω την συμπερίληψη αυτή. Τελικά προσπάθησα να έχω ευρύ φάσμα γεωγραφικών παραδειγμάτων ώστε να μην ε, αναφερόμαστε σε μία χώρα μόνο και ελπίζω η συμβαστική τροπολογία να το αντικατοπτρίζει αυτό. Όσον αφορά την παράγραφο 6 που ουσιαστικά έχει να κάνει με το πλαίσιο της ε, οικονομικής κάμψης ε, λόγω της οικονομικής κρίσης. Έχουμε εδώ το παράδειγμα του offshoring και μαζί με την κυρία Χάρκινς συμφωνήσαμε να μιλάμε για την αναλογικότητα όσον αφορά την ε, απώλεια θέσεων εργασία ε, και να έχουμε καλύτερη πρόσβαση στην αγορά για του ε, ευρωπαϊκού εμπόρου. Πιστεύω ότι αυτή είναι η ισορροπημένη προσέγγιση και μπορώ να την στηρίξω. Και τέλο, όσον αφορά την παράγραφο 7. Συγκεκριμένη παράγραφο για τις εμπορικές συμφωνίες όπου αναφερόμαστε στη διαδικασία του Heiligendamm, την οποία κίνησε η προηγούμενη Γερμανική Προεδρία η κυρία ε, ε, Ρέρνε, ε, η αγαπητή συνάδελφός μας, με την, οποία, την οποία ακολουθώ σε κάθε συνεδρίαση της σήμερα το απόγευμα, θα δω πού θα πάει μετά για να, για να πάω κι εγώ, την ενδιαφέραν πολύ τα όσα αναφορά ήθελε να συμπεριληφθούν τα όσα, όσα αφορούν τις επενδύσεις στη συνθήκη και έτσι καταλήξαμε στην βεβαστική τροπολογία 4. Δεν είχαμε πολύ χρόνο, δεν είμαι βέβαιος ε, δεδομένη της πίεσης του χρόνου ε, ότι είναι χρήσιμο να επαναλάβουμε τις συζητήσεις που είχαμε στο παρελθόν. Πολύ ευχαρίστω όμως θα απαντήσω σε ενδεχόμενες ερωτήσεις ή παρατηρήσεις ε, σχετικά με τις ε, προτάσεις τροπολογιών για την ε, γνωμοδοσία αυτή. Να πω στον κύριο Κάσλερ και στο ΕΛΚ ότι εκεί που προτείνεται διαγραφή, πολύ ευχαρίστως δέχτηκα τροπολογίες, αλλά το να διαγράφονται ολόκληρες παράγραφοι μου φαίνεται υπερβολικό. Θα ήθελα να σκεφτείτε μήπως μπορείτε να αποσύρετε τις τροπολογίες αυτές διότι κατά τα άλλα πιστεύω ότι έχουμε ένα πολύ οικοδομητικό και ισορροπημένο κείμενο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Merci beaucoup. Merci de ces amendements de compromis. Σα ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ για αυτέ τι συμβαστικέ τροπολογίε. Υπάρχουν <coughs> παρεμβάσει, παρατηρήσει επικρίσει, έπαινη, όχι τίποτα. Όλα αυτά μας αφήνουν να φανταστούμε ότι αύριο από τις 11 και μετά θα ψηφίσουμε υπό καλές συνθήκες. Ολοκληρώσαμε τις εργασίες μας για απόψε και σας εύχομαι καλό σας βράδυ.